Państwa, zaczynamy. Nie ma, rozumiem, uwag do porządku dziennego. Tłumaczenie mamy na 17 Λοιπόν, ξεκινάμε. Αν δεν έχουμε σχόλια για την μερίσια διάταξη, έχουμε διαμηνήσει 17 γλώσσες και η συνεδρίαση ε, μεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο. Υπάρχουν, ε, αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, μπορούμε να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της προηγούμενης ε, συνεδρίασης και χαιρόμαστε που έχουμε σήμερα μαζί μας τον Επίτροπο Χόγκαν που είναι υπεύθυνο για ε, θέματα αρμοδιότητάς μας. Είναι η οδηγία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές στη, στον τομέα των τροφίμων. Γιατί υπάρχουν σοβαρές ανισορροπίες στην αλυσίδα τροφίμων και χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια. Το Νοέμβριο του 2015 η Επιτροπή μας μαζί με την ΙΜΚΟ έκανε μια έκθεση ιδέας πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό με βάση τον ε, κανόνα 54 που έχει κοινή αρμοδιότητα. Ακριβώς για τις ε, θέμητες εμπορικές πρακτικές στην ε, αλυσίδα παροχής τροφίμων. Η κυρία Μαγκίνη ήταν η συγκήτριά μας. Στην έκθεση αυτή καλέσαμε ε, να υπάρξει νομοθεσία για το θέμα αυτό. Και επίσης στις 7 Ιουνίου 2016 υπήρξε ένα ψήφισμα του Κοινοβουλίου όπου το Κοινοβούλιο καλούσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει προτάσεις κατά αυτών των αθεμήτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα παροχής τροφίμων ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ένα δίκαιο εισόδημα για τους ε, γεωργούς, ε, ευρία επιλογή για τους καταναλωτές και διαφανεί σχέσεις μεταξύ των παραγωγών και διανομέων τροφίμων. Επίσης, δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα, Task Force για την Γεωργία, που υπέβαλε έκθεση τον περασμένο Νοέμβριο, όπου πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εισαγάγει ένα νομοθετικό πλαίσιο για τα θέματα αυτά, ούτως ώστε να υπάρξει μια εναρμονισμένη ελάχιστη βάση που να προβλέπει ποιες αθέμητες εμπορικές πρακτικές πρέπει να απογορευτούν και να υπάρξουν οι αναγκαίοι κανόνες για να λειτουργήσει αυτή η νομοθεσία. Υπάρχουν ε, κανόνες της Ένωσης, ε, ε, δηλαδή πρότεινε ότι θα μπορούσε να, υπάρξει, να υπάρξουν κανόνες της Ένωσης ή κανόνες των κρατών μελών οι κώδικες ε, δεοντολογίας. Και η πρόταση αυτή λοιπόν εγκρίθηκε από τους επιτρόπους, από το Σώμα των Επιτρόπων και με πολύ χαρά σήμερα καλωσορίζουμε τον Επίτροπο Χόγκαν για να μας παρουσιάσει αυτή την πρόταση. σε αυτή την ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Κατόπιν ε, βεβαίω ε, θα υπάρξουν ε, ερωτήσει, απαντήσει, αλλά πρώτα απ' όλα να μα κάνει την παρουσίαση του Επίτροπο, τον οποίο και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ για να αντιμετωπίσουμε σήμερα αυτό το θέμα τη τροφιμική αλυσίδα και των αθεμήτων πρακτικών και νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα που κάνουμε στο μακρύ ταξίδι για μια πιο δίκαιη και πιο λειτουργική ε, τροφιμική αλυσίδα. Βέβαια, το μεγαλύτερο τμήμα του ταξιδιού τώρα ανοίξει στο παρελθόν. Τώρα, με την δημοσίευση αυτή τη πρόταση βλέπουμε φως ε, στο τέλο του τούνελ. Σήμερα δείχνουμε ε, πώ λειτουργεί μια Ευρώπη που προστατεύει στον τομέα τη γεωργία και των τροφίμων. Και αποδεικνύουμε στου πολίτε μα ότι η συνεργασία σε ενωσιακό επίπεδο μπορεί να προσθέσει σαφώ αξία στην καθημερινότητά τους Ήθελα να έρθω ακριβώς εδώ στο Κοινοβούλιο, γιατί πολλά από τα μέλη σας έχουν παίξει σημαντικό ρόλο για να τεθεί αυτό το θέμα στην μέση συνένταξη εδώ και πολλά χρόνια. 19 χρόνια συγκεκριμένα. Ιδιαίτερα να αναφέρω την έκθεση τη Αντιπρόεδρου Μαγκίνε που τη βοήθησε ο κ. Δεκάστροπο τόσο καλά και τι γνωμοδοτήσει ΔΕΛΑΕ και τη στήριξη όλων των συντονιστών και όλων των μελών ε, του σώματό σα για την πολύ ισχυρή εντολή που έλαβε η Επιτροπή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να κάνουμε κάτι για το θέμα αυτό. Υπήρξε λοιπόν το 2017 ε, σαφές μήνυμα. Η, το ψήφισμά σας που ενεκρίθη τον Ιούνιο του 2016 τόνισε με πολύ σαφή και περιεκτικό τρόπο τι θέματα τίθενται και τις προκλήσεις για την διαμόρφωση πολιτικής. Είστε το προγεφύρωμα της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, εκλέγεστε άμεσα για να εκπροσωπήσετε τους πολίτες. Ακούτε λοιπόν πολύ καλά τη φωνή των καταναλωτών σε κάθε περιφέρεια. Και είναι εντυπωσιακό ότι πολλέ από τι ε, περιοχέ τη Υπέθρου που εκπροσωπείται έχουν εντοπίσει αυτό το, πρόγραμμα, το πρόβλημα. Συγγνώμη. Επίση, πρέπει να επενέσω την εργασία τη Σλοβακική Προεδρία στο δεύτερο εξάμεινο του 2016. Έτσι, είχαμε ομόφωνες, ε, ε ομόφωνα απορίσματα του Συμβουλίου. Και η Επιτροπή το 2016 δημιούργησε μια ειδική επιτροπή για τις ε, αγορές γεωργικών προϊόντων για να εκτιμήσει το ρόλο των ε, γεωργών στην ευρύτερη αυτή αλυσίδα και για να κάνει συστάσεις. Στη βάση αυτή η Επιτροπή έκανε μια αρχική μελέτη αντικτύπου και μια δημόσια διαβούλευση για τη βελτίωση αυτής της αλυσίδας το 2017 με βάση τη Διοργανική Συμφωνία για καλύτερες ρυθμιστικές διατάξεις. Και το αποτέλεσμα αυτής της διαβούλευσης μας βοήθησε να ε, εντοπίσουμε τις συγκεκριμένες αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Όπως ξέρουμε αυτές οι αθέμητες πρακτικές είναι πρακτικές μεταξύ επιχειρήσεων που δεν είναι σωστές εμπορικές πρακτικές και είναι κατά στην καλή πίστη και την ισότιμη αντιμετώπιση. Συνήθως επιβάλλονται μόνο μερός από τον ένα εμπορικό εταίρο στον άλλον. Η τροφιμική αλυσίδα είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες πρακτικές λόγω των μεγάλων διαφορών διαπραγματευτικής ισχύω. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση ενωσιακή που δημοσιεύθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο δείχνει ότι οι περισσότεροι που απάντησαν σε αυτή τη δημοσκόπηση, 88% θεωρούν ότι η ενίσχυση του ρόλου των γεωργών σε αυτή την αλυσίδα είναι πολύ σημαντικό. 99% αυτοί που απάντησαν στη δημόσια διαβούλευση το 17 για την, τον εξυγχρονισμό τη ε, ΚΑΜΑ, της ΚΓΠ συμφωνούν με την πρόταση ότι η βελτίωση τη θέση των γεωργών σε αυτή την αλυσίδα, ιδιαίτερη αντιμετώπιση αυτών των πρακτικών, θα έπρεπε να είναι στόχο τη κοινή γεωργική πολιτική. Φυσικά υπάρχουν και εθνικές πρωτοβουλίες που έδειξαν τον δρόμο. Ιδιαίτερα ο νόμος για την τροφινική αλυσίδα στην Ισπανία και ο επιδιαιτητής ε, για τα θέματα γεωργικών προϊόντων στον Ηνωμένο Βασίλειο. Αλλά, όπως το ψήφισμά σας λέει και το παραθέτω, ο κατακαιρματισμός της αγοράς από διαφορετικές εθνικές προοπτικές δεν επιτρέπει να αντιμετωπιστούν αυτές οι πρακτικές. Η λύση που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, μια νομοθεσία πλαίσιο σε ενωσιακό επίπεδο για να αντιμετωπιστούν αυτέ οι πρακτικέ και ούτω ώστε οι γεωργοί και οι καταναλωτέ να έχουν δυνατότητα να υποφεληθούν από δίκαιε πρακτικέ ε, αγοραπολισιών, τώρα θα γίνει πραγματικότητα. Για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Ε, Τέτοιε δράσει συζητούνται εδώ και πάνω από 19 χρόνια και τώρα επιτέλου έχουν γίνει πραγματικότητα. Προτείνουμε συγκεκριμένα και στοχευμένα μέτρα που θα έχουν αντίκτυπο στα πιο αδύνατα σημεία τη τροφιμική αλυσίδα. Γιατί μια αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή όσο ο πιο αδύναμο κρίκο τη. Οπότε αυτέ οι αλυσίδε, συγγνώμη, αυτέ οι ενέργειε θα ωφελήσουν του πάντε. Από το γεωργό μέχρι τον καταναλωτή. Οι ε, αθέμητε πρακτικέ που θα πρέπει να αγορευτούν είναι ε, ε, καθυστερημένε πληρωμέ για αναλώσιμα, ε, ακυρώσει τελευταία στιγμή των παραγγελιών, ε, μονομερεί ή αναδρομικέ αλλαγέ στα συμβόλαια και να υποχρεώνεται ο παραγωγός να πληρώσει για προϊόντα που δεν πουλήθηκαν ή τα οποία σάπησαν. Άλλες πρακτικές που θα επιτρέπονται μόνο αν υπάρχει σαφής συμφωνία μεταξύ των ε, ε, συμβαλωμένων είναι η εξής. Θα είναι, για παράδειγμα, ε, ο αγοραστής να επιστρέφει τα απόλυτα προϊόντα ή να επιβάλλει πληρωμές για να διατηρηθεί η συμφωνία πώλησης. Ένας ε, παραγωγό ο οποίο θα πρέπει να πληρώσει για τη διαφήμιση των προϊόντων που θα πουλήσει ε, το σούπερ μάρκετ. Και επίση προτείνουμε να υπάρχει ένα σώμα που να ελέγχει την εφαρμογή των κανόνων. Μια νομοθεσία αξίζει μόνο να μπορεί να εφαρμοστεί. Και αν υπάρξουν παραβάσει, το υπόφθηνο σώμα θα μπορεί να επιβάλλει όχι δυσανάλογε και αποτρεπτικέ ε, κυρώσει. Φυσικά πρέπει να έχει και ισχυρέ αρμοδιότητες αυτό το σώμα οποιοδήποτε κάνει ε, ε, αίτημα θα μπορεί να αντιμετωπιστεί το αίτημά του και θα αντιμετωπιστεί με συνθήκες ε, ανωνυμίας για να μην εκφοβίζεται κανένας. Αλλά φυσικά είμαστε μια ενότητα ίσων. Κανένας δεν έχει το μονοπόλιο της οφροσύνης. Γι' αυτό θα υπάρχει και ένας μηχανισμός συντονισμού μεταξύ αυτών των αρχών επιβολή για να ανταλλάσσονται ευέλικτε πρακτικέ. Η επικουρικότητα και η αναλογικότητα φυσικά είναι τα βασικά μα μελήματα. Άρα αυτά τα μέτρα συμπληρώνουν τα μέτρα που ήδη ισχύουν στα κράτη-μέλη και ο κώδικας ε, δεοντολογίας και του κώδικα δεοντολογίας για την εθελούσια ε, πρωτοβουλία για την ε, διατροφική αλυσίδα. Τα κράτη-μέλη μπορούν να λάβουν και συμπληρωματικά μέτρα. Και βεβαίω θα κάνουμε πρώτα απ' όλα μια πολύ καλή μελέτη αντικτύπου που θα υποβληθούν και τα δύο και το νομοθέτημα. Και η μελέτη αντικτύπου στι δύο συνομοθετικέ αρχέ. Είναι βεβαίω ε, πολύ φρέσκια αυτή η πρωτοβουλία, οπότε και στο μέλλον θα είμαι διαθέσιμο για να απαντήσω ερωτήσει. Ε, όταν θα έχετε δυνατότητα ακριβώ να μελετήσετε σε βάθο αυτή την πρωτοβουλία. Η ενίσχυση τη θέση ε, των παραγωγών στην τροφιμική αλυσίδα ήταν πάντα μεγάλη προτεραιότητα για μένα. Την ανέφερα εδώ και στην αρχική μου ακρόαση του 2014. Η συνεργασία των θεσμικών οργάνων, όπω απαιτούν οι πολίτε, επιτρέπει να επιτύχουμε πολλά. Μαζί έχουμε ήδη διευκολύνει τους ε, γεωργούς μέσω του όμνιμπους για να οργανώνονται και να διαπραγματεύονται για την πώληση των προϊόντων τους. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Τότε το όμνιμπους, το δεύτερο βήμα είναι η σημερινή πρόταση και το τρίτο βήμα θα είναι μια πρωτοβουλία για να βελτιωθεί η διαφάνεια των αγορών. Ε, ελπίζω να υποβάλω αυτή την πρόταση ακόμη φέτος. Καταλήγοντας, μια τροφιμική αλυσίδα που θα διακυβερνείται σωστά πρέπει να είναι ισότιμη. Η πρόταση είναι για δικαιοσύνη και για του Γεωργού σήμερα. Για να δώσουμε φωνή σε αυτού που δεν έχουν φωνή, που χωρί να φταίνει οι ίδιοι πολλές φορές είναι θύματα τη ε, αδύναμη διαπραγματευτική του θέση. Η αντιμετώπιση αυτών των αθέμητων πρακτικών είναι καλή βάση για περαιτέρω εργασία σε αυτόν τον τομέα και φυσικά βασίζουμε και στη δική σας ε, ε, συμβολή για να προχωρήσουμε περαιτέρω αυτή τη διαδικασία και τη στήριξή σα Σα ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πρόταση λοιπόν είναι επιτάπητος. Ο πρώτος που θα πάρει το λόγο είναι ο κ. Χάσλινγκ, γιατί οι πράσινοι έχουν ένα σεμινάριο για την κοινή γεωργική πολιτική σήμερα. Οργανώσαμε αυτή ε, την, εδώ τη συνεδρίαση αργότερα, αλλά εσείς θα χρειαστεί να φύγετε σύντομα, γι' αυτό και έχετε το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και όντω ε, αυτή τη ε, διάσκεψη της ομάδας την είχαμε οργανώσει εδώ και καιρό και η πρόσκληση του κ. Χόγκαν ήταν πρόσφατη. Και γι' αυτό λοιπόν σα ευχαριστούμε που μα δίνετε το λόγο πρώτα-πρώτα. Ευχαριστούμε, Επιτροπέ, για την πρωτοβουλία σα. Πήρε καιρό τελευταία στιγμή ε, στη θητεία προέκυψε η πρόταση, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι μια προσέγγιση. Όλα αυτά τα οποία αναφέρθηκαν ε, κατά τα θέμη των εμπορικών πρακτικών είναι πραγματικά Πράγματα που πρέπει να έχουν γίνει το και καιρό σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τι προθεσμίε ε, πληρωμή και όλα αυτά που χρειάζονται οι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όλα αυτά λοιπόν είναι καλά και ωραία. Αλλά ένα πρόβλημα δεν επιλύεται. Αυτό που αναφέρεται και στην έκθεση μακίνε. αυτή η ανισορροπία του τι μπορούν να κάνουν οι μικρέ επιχειρήσει ε, έναντι των μεγάλων μονοπωλίων. Έχουμε λοιπόν δυο-τρει εταιρείε στη Γερμανία που καθορίζουν την διατροφική αλυσίδα. Αυτή η δυσαναλογία λοιπόν είναι θέμα δικαιωμάτων καρτέλ. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε κάτι στο επίπεδο αυτό προκειμένου και οι μικροί πάροχοι, οι μικροί προμηθευτές, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μπορέσουν να έχουν τα δικαιώματά τους. Άρα, καλωσορίζω τα όσα αναφέρατε, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτελέσουν μία αυτά τα μέτρα. Το λέω αυτό ξεκάθαρα. Θα πρέπει να πάμε και παραπέρα. Και το είπαμε και σε όλες τις εκθέσεις. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι τα μονοπόλια σήμερα καθορίζουν τις ε, αλυσίδες ε, παρομήθειας τροφίμων στα καταστήματα και οι υπόλοιποι μικροί τρέχουν και δεν προβλέπουν. Το θέμα των προθεσμιών πληρωμής αποτελεί ένα ζήτημα. Το αναφέρατε. Αυτό τι δείχνει. Εντάξει, μπορούν να καταγγελθούν τα προβλήματα, αλλά στην τελική ανάλυση, τι σημαίνουν αυτές οι καταγγελίες, τι αλλαγές μπορούν να επιφέρουν, τι διαφορά μπορούν να σημειώσουν. Αυτό είναι το θέμα λοιπόν το οποίο με απασχολεί. Το πήραμε χθε το βράδυ το κείμενο και νομίζω ότι αναφέρονται 14 σημεία τα οποία όντω υποτίθεται ότι θα αλλάξουν κάτι στην κατάσταση. Ελπίζω και αναμένω από πλευρά της έκθεσής μας. Να ζητήσουμε να αλλάξουν σημαντικά στοιχεία. Να μπουν στο κείμενο και στοιχεία από την έκθεση Μακίνες για να ενισχύσουμε την έκθεση προκειμένου τελικά να σημαίνει και στην πράξη κάτι για τους μικρούς παραγωγούς. Όπως σας είπα δεν αναφέρει το βασικό πρόβλημα, δυστυχώ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που είναι η δυσαναλογία που επικρατεί με την παρουσία μονοπωλίων. Γιατί δεν το θέτει λοιπόν το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν το συζητά με την Επίτροπο Ανταγωνισμού. Αυτό είναι θέμα προσέγγιση. Και κατά δεύτερον, θα πρέπει να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε το θέμα των μονοπωλίων. Ευχαριστώ πολύ. Εκτό μικροφώνου, ο Πρόεδρο. Το λόγο έχει ο επόμενο ομιλητή. Euh, Μάλιστα. Ο κύριος Μποβέ, ευχαριστώ. Είναι, είναι κάτι που οδεύει προς σωστή κατεύθυνση, αλλά πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις. Καταρχάς, η διαφορά απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις ε, και τα μεγάλα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, τις μεγάλες γαλακτοκομικές εταιρείες που μπορούν να προσφέρουν πολλά διαφορετικά προϊόντα στη διαπραγμάτευση και τις, μεγάλες, τις μικρές μάλλον εκμεταλλεύσεις που έχουν λίγα προϊόντα γιατί η πίεση επ' αυτών είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι στις μεγάλες που αυτές εφόσον δεν συμφωνούν για μια τιμή μπορεί να το καλύψουν από μια άλλη. Οπότε μπορεί να υπάρχει μεγάλη ε, στρέβλωση λόγω της ε, διάσταση τη επιχείρηση. Αυτό είναι πρόβλημα και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό τι διαπραγματεύσει. Το δεύτερο πρόβλημα αφορά του παραγωγού. Έχουμε πολλέ μεγάλε επιχειρήσει. Θα σα αναφέρω τη Λακταλή τη Γαλλία, που σίγουρα γνωρίζετε πολύ καλά, που δεν παρουσιάζει ε, λογαριασμού, ε, ισολογισμού γιατί δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Αυτό σημαίνει πω οι παραγωγοί σήμερα δεν έχουν τη δυνατότητα διαπραγματεύση ε, με βάση το πραγματικό πραγματικότητα του κόστους που επιβάλλεται στους παραγωγούς. Οπότε έχουν πάρα πολύ δύσκολη, μεγάλη δυσκολία και σε αυτό το σημείο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έπρεπε να υπάρχει μια υποχρέωση διαφάνειας για τους λογαριασμούς και οι ε, επιχειρήσεις να μην μπορούν να κρυφτούν πίσω από την νομοθεσία κάθε κράτους για να μην υποβάλλουν τα στοιχεία που είναι το σημείο εκκίνησης για κάθε διαπραγμάτευση. Σας ευχαριστώ. Κυρία Χόιμπος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο για την πρόταση που μας υπέβαλε. Και εγώ πιστεύω ότι ήταν απαραίτητη. Αλλά και εγώ πιστεύω και ανέφερε ο κ. Μποβέ το παράδειγμα της Λακταλής ότι δεν κοιτάμε τι γίνεται μεταξύ μεταπηγητών και ε, σούπερ μάρκετ καλό και αυτό το στοιχείο, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε και το ρόλο των ε, γεωργών, των ε, μεταποιητών, έναντι, για παράδειγμα, των γαλακτοκομικών επιχειρήσεων. Στη Γερμανία υπάρχουν και πολλές ε, ενώσεις. Και αυτοί λοιπόν έχουν αγοραστική δύναμη και αντιμετωπίζουν και οδηγούν κάπως τον καταναλωτή. Ύστερα, έχω και κάποιες αμφιβολίες. Γιατί αναφέρεται ένα κατάλογο. Ένα κατάλογο αθέμητων εμπορικών πρακτικών. Και είμαι σχετικά βέβαιη ότι οι δικηγόροι των ομίλων θα κάτσουν να κοιτάξουν τον κατάλογο αυτό και να δουν πώς θα μπορέσουν να ξεφύγουν από όλα τα στοιχεία αυτά. Το θέμα λοιπόν που θα θέλω να θέξω είναι το εξή. Θα παραμείνει κλειστός αυτός ο κατάλογος ή αν στη συνέχεια ανακύψουν και άλλες αφέμητες εμπορικές πρακτικές θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο κατάλογο αυτό. Προκειμένου να μην ε, αρχίσουν και τους ε, πατάν τους γεωργούς με άλλο τρόπο απλά από ό,τι τους πατάν μέχρι τώρα. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να γίνει, να είναι ανοιχτός ο κατάλογος αυτός και το δίκαιο του ανταγωνισμού το ανέφερε και ο κύριος Χόισλεν. Υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση να τροποποιηθεί το δίκαιο ανταγωνισμού γιατί θεωρώ ότι αυτό αποτελεί την αιτία του προβλήματος. Ευχαριστώ πολύ και να δώσουμε το λόγο στον Επίτροπο για να απαντήσει στις πρώτες αυτές ερωτήσεις. Γιατί κάποιοι θα φύγουν από εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Πράσινου Κόμματος ε, για τα σχόλια τους. Κανονικά θα πρέπει να ανησυχώ που συμφωνείτε μαζί μου σε σχέση με αυτή την πρόταση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτά που είπατε ε, είναι αυτά που κάνουμε σε αυτή την νομοθεσία, αλλά μάλλον δεν είχατε την ευκαιρία να το μελετήσετε ακόμα. Ασχολούμαστε και αντιμετωπίζουμε όλους τους φορείς, όχι μόνο τον Γεωργό και τον Λιανοπολτή. Ε, και έπειτα είπατε ότι ο κατάλογος που έχω είναι μια πρόταση. Μετά οι συνομοθέτες ε, ε, θα το βελτιώσουν ή θα το αλλάξουν, εν πάση περιπτώσει, αφού ξέρετε έτσι πάει το πράγμα. Ε, και μετά έχουμε και τρία χρόνια για να χρησιμοποιήσουμε τον μηχανισμό αναθεώρησης. Ε, υπάρχουν λοιπόν όλα αυτά, έχουν προβλεφθεί. Η βασική ε, προσέγγιση λοιπόν εδώ κύριε Μποβέ και κύριε Χόσλινγκ είναι ακριβώς να στοχεύσουμε εκεί που έγινε το πρόβλημα, όπου δηλαδή ο Γεωργός ε, σαφώς έχει δυσκολευτεί σε σχέση με το δικό του μερίδιο της δράσης και όλους τους φορείς της διατροφημικής αλυσίδας. Η λακταλής μπορεί να καλυφθεί από την εθνική νομοθεσία αλλά και από νομοθεσία που θα υποβάλουμε αργότερα φέτος για τη διαφάνεια της αγοράς. Προσπαθούμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους παραγωγούς να έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική εξουσία και ισχύ ε, ως τμήμα της τροφιμικής αλυσίδας, να τους ενισχύσουμε. Έχουμε αυτή την πρωτοβουλία για τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές και ε, θα καταθέσουμε και νομοθεσία για τη διαφάνεια της αγοράς αργότερα. Επίσης έχουμε θεσπίσει παρατηρητήρια των αγορών σε κάθε τομέα, του, ε, τομέα της υγείας και των τροφίμων, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν το πράσιν, τους πράσινους που αναφέρατε όλα τα προβλήματα, αλλά και τις, έτσι μου δίνετε την ευκαιρία να αναφέρω τις λύσεις που περιλαμβάνονται στην πρόταση. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τέσσα, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω για τον Επίτροπο που μας κατέθεσε σήμερα την πρόταση αυτή και να ευχαριστήσω και την κυρία Μαγκίνες η οποία εργάστηκε πολύ σκληρά. Χαίρομαι που έχουμε λοιπόν αυτή την πρόταση μπροστά μας και τώρα είναι στα χέρια του Κοινοβουλίου το να εργαστεί γρήγορα και να βελτιώσει την πρόταση. Να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κύριος Χόισλινγκ. Είναι καλή η πρόταση, αλλά πρέπει να διευρυνθεί. Πρέπει να ενισχυθεί για να υπάρξει και αποτέλεσμα. Το θέμα λοιπόν είναι να αλλάξει το δίκαιο ανταγωνισμού. Και κύριε Επιτροπέ, είπατε και δικαίω ότι είναι η πρώτη φορά στο πλαίσιο αυτό στον τομέα αυτό τονίζω, γιατί το 2004 ήρθα εδώ στο Κοινοβούλιο, το 2005 λοιπόν κάναμε μια πολύ μαζική παρέμβαση σε ό,τι αφορά τους ε, ομίλους, σε ό,τι αφορά την περιαγωγή. Αν δεν είχαμε ξεκινήσει λοιπόν τότε τη διαδικασία αυτή, ακόμα roaming θα πληρώνουν οι πολίτες μας. Οι άδικες λοιπόν αυτές πρακτικές των ομίλων τερματίστηκαν. Και είναι αυτό φυσικά προ όφελο των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά έχουμε πετύχει. Άρα, έχετε συμπεριλάβει διάφορα στοιχεία τα οποία πάντα ζητούσα σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, ε, σταθερή προθεσμία ε, για πληρωμέ, ε, τέλη καταχώρηση σας ευχαριστώ λοιπόν που η Επιτροπή αυτή συμπεριέλαβε τα στοιχεία αυτά και που μας κατέθεσε την πρόταση για να εργαστούμε από αυτή στο Κοινοβούλιο. Έκαναν διάφορες συζητήσεις και με διάφορες ενώσεις και με μεταποιητές και αυτό που άκουσα ομόφωνα από όλους είναι ότι αντιμετωπίζουν τεράστιε πιέσει από τους μεγάλους ομίλους και δεν μπορούν να το καταγγείλουν αυτό γιατί πολύ απλά φοβούνται του μεγάλου ομίλους. Θα πρέπει να σπάσουμε λοιπόν αυτόν τον κύκλο, το φαύλο κύκλο και θα πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν και του γεωργού, αλλά και τι εταιρείε μεταποίηση. Ξέρω μια επιχειρήση με δισεκατομμύρια κύκλο εργασιών και ακόμα και αυτή η ε, επιχείρηση, σα πληροφορώ ότι αισθάνεται τεράστια πίεση και ότι την εκβιάζουν ουσιαστικά οι μεγάλοι όμιλοι. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λοιπόν, ε, Επίτροπε, και να είστε σίγουρο ότι η ομάδα μου θα εργαστεί πάρα πολύ σκληρά προκειμένου να πετύχουμε μέσα σε θετία αυτή καλά αποτελέσματα. Και ξέρω ότι αυτά που σα είπαμε ενδεχομένω να μην ε, συναρπάσουμε την Επίτροπο την Αρμόδια για τον ανταγωνισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπολογίζετε στην υποστήριξή μα. Ο κύριο Αγνιό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για αυτή την πρόταση οδηγίας. Ευχαριστώ για την παρουσίαση που μας κάνετε σήμερα αλλά και για τα όσα είπατε όσον αφορά την μέρη σας στο... για το άνοιγμα που κάνετε για αυτό το βασικό κείμενο το οποίο θα μπορέσουμε να δουλέψουμε. όντω δεν προλάβαμε παρά να, τρέξουμε το κείμενο, αλλά ε, πρόκειται για μια καλή πρωτοβουλία. Ε, εδώ και καιρό χρειαζόμαστε μια τέτοια πρωτοβουλία. Ε, τα προβλήματα της τροφιμικής αλυσίδας δεν είναι καινούρια και γι' αυτό και χαιρόμαστε για αυτήν εδώ την πρωτοβουλία. Τα κράτη λοιπόν θα πρέπει να μπορούν να ενεργήσουν για να επιβάλλουν το σεβασμό των συμβάσεων. Θα πρέπει να δούμε όμως και ποιο είναι το αίτιο της έλλειψης ισορροπίας και να προσφέρουμε άμεσα και έμεσα ε, ε, Άμεσε και έμεσε λύσεις. Τώρα, πρακτική ε, αθέμητη, ε, δεν κάνουμε να σας πω τίποτα σε σχέση με τη συγκέντρωση στη μεγάλα ε, σούπερ μάρκετ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, όχι μόνο για την αγροτροφημική αλυσίδα, αλλά και για τις μεγάλες προμήθειες. Αυτό δημιουργείται πρόβλημα. Η το τελευταίο παράδειγμα, δηλαδή η εξαγορά της Μονοσάντο από την Πάγιαν δεν μπορεί παρά να μας ανησυχεί. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και είναι δική μας ευθύνη να προστατεύσουμε μέσω της νομοθεσίας τόσο τους καταναλωτές όσο και τους γεωργούς. Και αυτό ακριβώς σας λέμε εδώ, απέναντι σε αυτά τα μεγάλα ολιγοπόλια. Εξάλλου σε ένα άλλο επίπεδο και δεν είναι το ίδιο θέμα, στο ίδιο επίπεδο μάλλον, είναι το θέμα των σημάτων των διανομέων που θα πρέπει να εμφανίζεται σε αυτή την οδηγία και δεν το έχω δει εγώ εδώ. Για μένα αυτό είναι το χαρακτηριστικό της ε, οικονομικής κυριαρχίας των μεγάλων ε, εταιριών διανομής, γιατί δεν δίνονται έτσι απαραίτητες πληροφορίες πληροφορίες ε, ε, ε, στους καταναλωτές. Τέλος, έχω να πω και κάτι για την ουδετερότητα του ίντερνετ. συζητάμε, αλλά θα πρέπει να συζητήσουμε και για την ουδετερότητα των μεγάλων διανομέων, γιατί έχουν τεράστια ισχύ για το τροφιμικό μας σύστημα. Ε, η καταπολέμηση των ε, θέμετων πρακτικών θα πρέπει να οδηγήσει και στα δικαιώματα υπεργολαβία στον τομέα των αγροτροφημικών. Αυτές είναι οι πρώτες μου παρατηρήσεις, αφού όπως σας είπα διάβασα βιαστικά την πρότασή σας, ε, εξάλλου θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Κυρία, Κυρία Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίζω ιδιαίτερως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε τη θέση των αγιοργών στην διατροφική αλυσίδα. Γιατί οι αγρότες μας δεν παίρνουν πάντα τις σωστές τιμές και σίγουρα δεν παίρνουν και τη σωστή μεταχείριση. Και φυσικά η διαδικασία μέχρι το σούπερ μάρκετ, μάλλον τελικά ωφελούνται άλλοι φορές. Αλλά φυσικά οι μεταπίτες δεν μπορούσαν να βγάλουν κέρδος αν δεν υπήρχαν οι αγρότες. Αναφέρατε το θέμα της επιδετησίας για τα τρόφιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, νομίζω ότι αποτελεί ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για να δείξουμε πού έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στα θέματα αυτά. Εγώ τον έχω τον κώδικα και τη σχετική έκθεση σε ό,τι αφορά την τελευταία του δημοσίευση. Κοιτώντας λοιπόν πώς έχει η κατάσταση, όταν η Κριστίνα ανέλαβε τα καθήκοντα αυτά, υπήρχαν ε, αγρότε οι οποίοι επιβαρύνονταν υπερβολικά για τη συσκευασία, για παράδειγμα, για τις παλέτες, ε, για τα κασόνια από το σούπερ μάρκετ στα οποία ε, προμήθευαν τα αγαθά του. Υπερβολική λοιπόν χρέωση και μία από τις πιο ακραίε περιπτώσει ήταν η εξή. Αν ένα καταναλωτή, για παράδειγμα, γράψει μια καταγγελία για ένα προϊόν, τελικά το σούπερ το φορτώνει αυτό στον ε, αγρότη. Αλλά αυτό ακριβώ κάνουν όταν ο καταναλωτής γράφει... Ε, ένα γράμμα καταγγελία για το πόσο καλό ήταν ένα προϊόν. Άρα τελικά ο αγρότη καταλήγει να ζητά στον καταναλωτή να μην γράφει ποτέ και να λέει για παράδειγμα τι ωραία που ήταν τα του. Αυτό που είναι θερδικό είναι πόσο ο αριθμό των καταγγελιών από πλευράς των γεωργών έχει μειωθεί το τελευταίο έτος για υπερβολική επιβάρυνση λιανική σε ό,τι αφορά ε, εκστρατείες ε, design από 22% σε 0%. Αυτό προφανώς είναι θαρρυντικό και με ικανοποιεί. Η νομική βάση του μέτρων αυτών σίγουρα θα πρέπει να είναι το άρθρο 43 και εμείς θα πρέπει να, είμαστε η κινητήριος δύναμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επίτροπε, η κυρία Μιούλερ, να σας ευχαριστήσω για την υποβολή μιας οδηγίας και όχι κανονισμού, γιατί πιστεύω ότι μια οδηγία στην προκειμένη περίπτωση αποτελεί τη σωστή λύση. Έχουμε τους βασικούς κανόνες από πλευράς της Ευρώπης και τα κρατημέλη θα έχουν τη μετότητα να τα δημορφώσουν αυτά όπως επιθυμούν. Γνωρίζουμε φυσικά ότι στα κρατημέλη επικρατούν διαφορετικά δικαιώματα σε ό,τι αφορά τα καρτέλ, αλλά νομίζω ότι και στη Γερμανία αντιμετωπίζουμε προβλήματα στα σύνορα. Ω τώρα δεν αντιμετωπίζονταν το θέμα αυτό σε εθνικό επίπεδο, γιατί το θέμα των καρτέλ έβαζε πάντα στο επίκεντρο των καταναλωτή ω τώρα και όχι ιδιαίτερα τον παραγωγό και τον μεταποιητή στην ε, διατροφική αλυσίδα. Είναι λοιπόν σωστό που γίνεται αυτή η πρόταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι δυνατότητε ε, αλλαγή για τις 30 ημέρες και δικαίωμα επιστροφή κτλ. Είναι καλά στοιχεία αυτά. Αυτό που μου λείπει ωστόσο είναι κάποια στοιχεία τα οποία έχουμε υπερψηφίσει στην έκθεση της κυρίας Μαγκίνης. Ήμουν και συνεισηγήτρια. Και αυτό που θα πρέπει σίγουρα να αναφέρουμε είναι τη δυνατότητα αυτή που ανοίξαμε στην Omnibus σε ό,τι αφορά την κοινή α, τάξη αγοράς. Αυτά θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε λοιπόν. Και φυσικά συνειδητοποιώ ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο φυσικά είναι το δίκαιο ανταγωνισμού μαζί με τα εθνικά δικαιώματα των καρτέλ. Αλλά νομίζω ότι ως προσέγγιση είναι η σωστή. Θέλουμε προφανώς και εμείς να εργαστούμε γρήγορα και αποτελεσματικά προκειμένου να είναι πιο σωστή η κατάσταση για τους αγρότες. Οι καταναλωτές στην Ευρώπη ε, είναι αυτοί που έχουν τα πιο πολλά πλεονεκτήματα. Αν τελικά καταφέρουμε να παράγουμε τα καλύτερα τρόφιμα. Thank Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις, Επίτροπε. Είναι καλά νέα Όπω είπαν και άλλοι, όμω ε, ο διάβολο κρύβεται στι λεπτομέρειε Για το πού θα καταλήξουμε θα δούμε. Πάντως σίγουρα είναι μια καλή αρχή. Κάτι που σίγουρα πρέπει να αλλάξουμε αν θέλουμε ο κόσμος να συνεχίσει να καλλιεργεί τη γη είναι να μπορούν να έχουν... Να, να πληρώνονται αντίστοιχα με την δουλειά που κάνουν. Και όσον αφορά τις ε, δίκαιες ε, επιδοτήσεις ε, άκουσα θετικές ιδέες ότι είναι δηλαδή θετικό το πώς θα πληρώνεται ο κόσμος, δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν 30 χρόνια. Ε, ε, αν όλα αυτά καρποφορήσουν, μάλλον θα μπορέσει ο κόσμος να παραμείνει στη γεωργία. Πράγματα τα οποία α, είναι, όπως ε, οι καθυστερημένες πληρωμές, πράγματα τα οποία έχουν σχεδιαστεί να συγχύσουν τους γεωργούς και να τους βάλουν στη θέση τους, μας κάνουν να τους κάνουν να αισθάνονται σαν να είναι ο Δαβίδ απέναντι στον Γολιάθ. Ελπίζω λοιπόν πως αυτή τη φορά έχουμε κάνει μια προσπάθεια ε, να προχωρήσουμε, να, να, εξισορροπήσουμε κάποιο την κατάσταση. Ε, όπως είπα όμως θα πρέπει να διαβάσουμε όλες τις λεπτομέρειες. Και για να πιαστώ από αυτό που είπε ο τελευταίο ομιλητής, διερωτώ με γιατί πήγαμε από το μηχανισμό που έχουμε σε μια οδηγία αντί για έναν ε, ε, κανονισμό. Η κυρία Μίλλερ εξήγησε πως ίσως είναι αυτό ευκολότερο να λειτουργήσει σε εθνικό επίπεδο. Εσείς όμως ε, με ποιο σκεπτικό το προτείνατε, γιατί παλιότερα έχετε πει ότι η κατακαιρματισμένη νομοθεσία που ήδη ισχύει δεν είναι αποτελεσματική. Γιατί λοιπόν να προτείνετε οδηγία αντί για κανονισμό. Δεν λέγω ποιο, δεν κρίνω ότι είναι το καλύτερο, απλά είμαι περίεργος να καταλάβω με ποια λογική ε, και πιο σκεπτικό ε, κάνατε αυτή την πρόταση. Πάντως μπράβο σας για την ώρα και νομίζω ποτέ δεν με ακούσατε να λέω τέτοιο πράγμα. Σας ευχαριστώ που συμφωνείτε μαζί μου επιτέλους, λέει ο Επίτροπος. Ευχαριστώ. Θα διαπιστώνετε από τα χαμόγελα εδώ στην αίθουσα ότι ο συνάδελφος Φλάνναγκαν μισοευχαρίστησε τον Επίτροπο, που πράγμα που δεν έχει ξανασυμβεί. Ε, όμως ε, ε, κομψά τα είπατε, αλλά αυτό που με ανησυχεί είναι ότι μήπως αυτή η δραστηριότητα της Ένωσης θα μπορούσε να υποβαθμίσει τον ε, το, το, το δικό μας, ε, τη δική μας κατάσταση, γιατί θα γίνει το Brexit, αλλά θα υπάρχει μια περίοδο που η Βρετανία στην ουσία θα στέκεται μόνη της και πιθανότητα υπάρχει μεγάλα καταστήματα, μεγάλη διανομή να μην ε, λειτουργήσουν καλά. Θα περιμένουν να δουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία για να δουν τι θα κάνουν. Εμένα με ανησυχεί αυτό. Εμείς έχουμε προδεύσει κάπως το Ηνωμένο Βασίλειο και πραγματικά δεν θα ήθελα να υποβαθμιστεί. Θα ήθελα να ακούσω και από τον Επίτροπο τι θα κάνει με τις τιμωρίες. Πώς θα τιμωρήσετε τα σούπερ μάρκετ ή μήπως θα γίνει ένα δικαστήριο, ε, μάλλον δίκες που θα ε, τραβάνε για χρόνια χωρίς να δίνετε μια λύση Επίση υπάρχει αυτό το δίλημα. Ο καταναλωτή πάλι θα πληρώσει την ύφη, θα πληρώνει όλο και περισσότερο στο σούπερ μάρκετ και αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Και κάτι ακόμα στο Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε πρόβλημα είναι το υποχρεωτικό συνταξιδοτικό για τους ε, εργοζόμενους όπου η παραγωγή, η υγειοργή θα πρέπει να πληρώνουν για ε, τη σύνταξη των εργαζομένων τους και τα σούπερ μάρκετ θα απασχολούν πολύ κόσμο όλοι αυτοί και τα σούπερ μάρκετ προσπαθούν να ε, καταφέρουν να επιδοτηθούν τα συνταξιδοτικά αυτά επιπλέον χρήματα, οι συνταξιδοτικές συνεισφορές από τους ε, προμηθευτές τους, ε, που και αυτοί πληρώνουν τις συντάξεις των δικών τους ε, υπαλλήλων. Τώρα, ένας γαλακτοπαραγωγός που έχει 70 γελάδες και μπορεί να παράγει γάλα, βούτυρο κτλ. Ε, μπορεί τώρα να λειτουργήσει καλύτερα με 500 αγελάδες. Ο κύριος Σουπόζο, ευχαριστώ Επιτροπέ. Ό,τι μας επιτρέψει επιτρέπει μάλλον να περιοριστεί η αυθέτη δύναμη ισχύς των μεγάλων δομών θα βελτιώσει τη ζωή των γεωργών και των κτηνοτρόφων. Ε, όσο γίνεται πιο χαμηλές τιμές στους καταναλωτές ε, είναι ο στόχος, ενώ οι ίδιοι καταναλωτές είναι έτοιμοι να πληρώσουν κάτι παραπάνω για ποιοτικά προϊόντα και να μπορέσει έτσι και ο παραγωγός να έχει πιο δικές τιμές. Γι' αυτό και βλέπουμε και την επιτυχία των εμπορικών δομών που τις διαχειρίζονται οι παραγωγοί χωρίς ενδιάμεσος Δυστυχώς οι άμεσες πωλήσει ε, είναι επιτυχής αλλά είναι δύσκολο ε, κανείς να έχει πρόσβαση γιατί χρειάζονται αρκετές επενδύσεις. Διαπιστώνουμε εδώ μια μορφή υποκρισίας. Όταν καταγγέλουμε τις εμπορικές αθέμητες πρακτικές ε, που ενώ τις εφαρμόζουμε σε διεθνές επίπεδο φαίνεται υποκρισία. Αυτό συμβαίνει όταν διαπραγματευόμαστε συνθήκες με την Μερκοσούρα, ας πούμε, που τις απορρίπτει ο επαγγελματικό τομέας γιατί πρόκειται για θέμα τον ανταγωνισμού. Κύριε Πίτροπε, προβλέπετε να σταματήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις για, το, για τη Μερκοσούρ που ομόφωνα έχουν απορριφθεί και θεωρούνται επικίνδυνες για τη γεωργία ε, και για την ασφάλεια των τροφίμων. Ευχαριστώ. δώσουμε το λόγο στον για να απαντήσει. Ευχαριστώ όλους τους συντονιστές που εξέφρασαν ε, τις απόψεις τους. Ε, μια αρχική άποψη βέβαια. Ο κύριος Ντάις έχει δίκιο. Δεν πέρασε εύκολα από την Επιτροπή αυτή η πρόταση. Με προσεκτικό τρόπο είπατε ότι δεν συμφωνούν όλοι οι Επίτροποι με τη δική μου γνώμη γι' αυτό. Και φυσικό ότι ε, τα θέματα της σχετικής ισχύω του καθενός και του ανταγωνισμού είναι βασικά. Ε, θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω όλους τους επιτρόπους που τελικά έχουμε μια πρόταση υπάρχει στήριξη για αυτή την προσπάθεια. Βεβαίω η πρόταση αυτή αφορά μόνο τα γεωργικά προϊόντα, τα γεωργικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται για τρόφιμα. Ελπίζω βεβαίω να συμμετάσχετε στη δουλειά και για περαιτέρω προτάσει και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε για να γίνει κάτι τέτοιο. Κύριε Ανδρέου, κάντε δύο παρατηρήσεις. Η πρόταση αυτή αφορά τις αθέμητες εμπορικές πρακτικές. Ξέρω ότι θα υπάρξουν ε, θέματα για το πεδίο εφαρμογής, αλλά τέτοια θέματα μπορούν να αφορούν την DG Grow με διαφορετικές νομικές δυνατότητες. Αλλά όλες οι σχέσεις μεταξύ των γεωργών και των μικρομεσαίων από τη μία και των μεγάλων μεταποιητών και διανομέων και ελιανεμπόρων από την άλλη μεριά καλύπτονται αυτή την πρόταση. Αυτή η οδηγία καλύπτει και τις διαμεθοριακές ε, δοσοληψίες. Και επίσης και τις σχέσεις με ε, παραγωγούς από τρίτες χώρες για να μην υπάρξει ε, καμία δυνατότητα κατάχρησης. Ευχαριστώ την κυρία Μαγκίνες. Ξέρω πόσο έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό και γενικά με το θέμα αυτού του επιδιαιτητή για τα τρόφιμα και τα χανικά ξέρω ότι αυτή η πρόταση έχει βοηθήσει το Ηνωμένο Βασίλειο. Πολύ θα ήθελα να μου στείλετε την ε, πρόσφατη ετήσια έκθεση αυτού του επιδιαιτητή γιατί μας δίνει στοιχεία για να δούμε τι ακριβώς λειτουργεί σωστά και στην Ισπανία. Υπάρχει ένας ε, επίσης νόμος για το τρόφιμα αλλά αυτές οι δύο χώρες είναι αυτές ε, που ε, μελετήσαμε πριν διατυπώσουμε την πρόταση. Ευχαριστώ κυρία Μαγκίνες για, για το ενδιαφέρον σας λοιπόν. Ο κύριος Μόρε και ο κύριος Φλάναγκαν ασχολήθηκαν με τα θέματα και ο κύριος Άγνερ. Γιατί οδηγία ρώτησαν και όχι κανονισμός. Εγώ νομίζω ότι η πρόταση αυτή είναι συμπληρωματική αυτών που συμβαίνουν στις χώρες μέλη και επίσης συμπληρωματική της πρωτοβουλίας για την ε, αλυσίδα παροχής τροφίμων. Και βεβαίως, αν ε, ε, προτείνει κανεί οδηγία, τότε τονίζουμε περισσότερο την επικουρικότητα. Κάποιες χώρες είναι πιο προωθημένε από άλλες και θέλουμε αυτό να αντανακλάται στην οδηγία μας, να υπάρχει μια σωστή ισορροπία. Γι' αυτό λοιπόν τελικά προτείνουμε οδηγία. Βεβαίως πρέπει να γίνει γνωστότερο το Omnibus, όπως είπαν και ο κύριος Δεκάστρο και άλλοι, και θα το κάνουμε τους επόμενους μήνες για να καταλάβουμε ότι είναι μια σταδιακή αλλαγή. Υπάρχει το Omnibus που ενισχύει τη θέση των παραγωγών μέσω των συνεταιρισμών και έχουμε επιτύχει πολλά με την ε, πολύ αξιόλογη ε, βοήθειά σας. Έχουμε επίσης αυτή την πρόταση τώρα, έχουμε τα παρατηρία των αγορών και θα προτείνουμε και περαιτέρω μέτρα για την διαφάνεια των αγορών. Άρα είναι ένα, μια δέσμη μέτρων, αλλά συμφωνώ ότι το Omnibus πρέπει να γίνει ευρύτερα γνωστό. Κύριε Φλάναγκαν, μα τι να πω. Χαίρομαι που επιτέλους ε, είδατε το φως ε, της δικαιοσύνης και με στηρίζετε. Ε, σας πήρε κάποιο χρόνο. Τρεις χρόνια είστε ευρωβουλευτής. Α, τέλος πάντων. Α, σχεδόν τέσσερα. Κύριε Άγγινιο, πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Τι πρόστιμα, πώς θα επιβληθεί η οδηγία. Η οδηγία αυτή δεν θα έχει έννοια εάν δεν εφαρμοστεί σωστά. Γι' αυτό είπαμε ότι θα υπάρχουν αυτές οι αρμόδιες αρχές με ουσιώδεις αρμοδιότητες, με δόντια. Αυτός ο σκύλος φύλαξ θα έχει δόντια. Κάθε χρόνο θα συναντιούνται όλες οι διάφορες ε, αρμόδιες αρχές στα κράτη-μέλη για να δούνε πώς έχει εφαρμοστεί αυτή η οδηγία δεν θέλουμε μόνο συντονισμένη άποψη για την ε, εφαρμογή της και τα πρόστιμα, αλλά θέλουμε να μελετήσουμε προσεκτικά την εφαρμογή της, να δούμε ποιες είναι οι βέλτιστες πρακτικές που μπορούν κατόπιν να ανταλλαγούν. Νομίζω ότι θα συμφωνούσατε ότι υπάρχει και επικουρικότητα. Μα υπάρχουν ήδη ρυθμίσεις στα κράτη-μέλη. Θέλουμε απλώς να τις συμπληρώσουμε, όχι να τις αντικαταστήσουμε. Αν τα κράτη-μέλη λοιπόν είναι σε καλύτερη θέση για να εφαρμόσουν τα πρόστιμα και τις κυρώσεις που ήδη υπάρχουν. Και έχουμε αυτό το παράδειγμα μέσω αυτού του επιδιαιτητή ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί διάφορες μεγάλες εταιρείες λόγω της εργασίας αυτής της αρχής έχουν συμμορφωθεί. Αυτό θα μπορούσε, με βάση λοιπόν αυτή τη βέλτιστη πρακτική, να επαναληφθεί και σε άλλες χώρες της Ένωσης. Και ξέρετε, οι επικρίσεις ε, που γίνονται ότι δηλαδή θα θαρδάρουμε τους καναλωτές με αυτές τις προτάσεις, με αυτές τις επικρίσεις από αυτούς που δεν θέλουν καμία αλλαγή. Οποτεδήποτε εφαρμόστηκαν τέτοιες αλλαγές, δεν έχουμε καμία ένδειξη αύξησης των τιμών καταναλωτή και όλες οι οργανώσεις των καταναλωτών που υπέβαλαν στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης τις απόψεις τους, στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Δεν νομίζω λοιπόν ότι οι οργανώσεις των καταναλωτών ε, στρέφονται κατά των συμφερόντων των μελών του. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δεν θα υπάρξει καμία αύξηση των τιμών καταναλωτή. Δημιουργεί ισότιμες συνθήκες ανταγωνισμού στην ε, εσωτερική αγορά και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Όχι μόνο με αυτό το νομοθέτημα, αλλά γενικότερα και με άλλα νομοθετήματα για την κοινή πολιτική. Είναι μια προσπάθεια να βοηθήσουμε τους πολίτες μας. Και αυτή είναι απάντηση και στο ερώτημα του κυρίου Λουαζό. Το ρόλο του καταναλωτή. Πώς θα φυγεί. Κατά τη διαδικασία της διαβούλευσης όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς είπαν ότι δεν νομίζουν ότι θα υπάρξει αύξηση των τιμών και για το Μερκοσούρ. Να τα πούμε άλλη μέρα αυτά. Λοιπόν, τώρα για μισό λεπτό οι επόμενοι ομιλητέ. Και πρώτα απ' όλα ο κύριο Ντεκάστρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ αγαπητέ Επίτροπε. Πιστεύω πως εδώ περιέχονται όλα τα συστατικά για να, έχουμε, να κάνουμε σωστή δουλειά. Και θυμήθηκα και αυτή είναι μια αρχική, πολύ σημαντική ε, πτυχή αρχικά. Η νομική βάση είναι μια νομική βάση που επιβάλλει ε, τούτη εδώ η Επιτροπή να έχει την ε, επί της ουσίας αρμοδιότητα. Και αυτό φυσικά πρέπει να το υπερασπιστούμε γιατί άλλες επιτροπές εδώ στο Κοινοβούλιο θα ήθελαν πολύ να, να γίνουν αρμόδιες από της ουσίας. Η νομική βάση μας θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε αυτή την μάχη. Όπως ε, ξέρετε, τότε η Επιτροπή, ε, ε, η Επιτροπή μας έχει κάνει σημαντική δουλειά για το Omnibus και σας ευχαριστώ που το αναφέρατε. Ήταν το πρώτο τμήμα της εργασίας της ειδική Task Force, γιατί έτσι προσπαθήσαμε να κάνουμε πιο δυσχυρές τις οργανώσεις των Γεωργών και δεν αποφύγαμε μια αντιπαράθεση με άλλες γενικές διευθύνσεις. Πιστεύω πως ήταν μια, ένα, ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα αυτή η αντιπαράθεση με την Γενική Διεύθυνση του Ανταγωνισμού. Αυτή η νέα πρόκληση λοιπόν με αυτή την οδηγία εδώ βέβαια μας ε, τοποθετεί στις ίδιες συνθήκες αλλά έχουμε ήδη αυτή την εμπειρία. Μια εμπειρία που μεταξύ άλλων έχουμε χρησιμοποιήσει στην Επιτροπή μας με τη δουλειά που έχει κάνει ήδη η Μαριάννα Μαγκίνες ε, μπήκαν στη σειρά διάφορα επιχειρήματα που αποσαφήνισαν τις θέμητες ε, πρακτικές στο εσωτερικό του τομέα αυτό, αλλά γνωρίζουμε πως υπάρχουν πάνω από 20 εθνικές νομοθεσίες, ορισμένες εξ αυτών πολύ ενδιαφέρουσες. Σίγουρα η ισπανική εμπειρία και η ε, αγγλική εμπειρία θα μας βοηθήσουν και θα μας κατευθύνουν και η εργασία εναρμόνισης με μία ε, ρύθμιση πλαίσιο που όμως θέλω να υπογραμμίσω που θα πρέπει να ορίζει ελάχιστε προδιαγραφέ, γιατί αυτό ε, περιλαμβάνεται και στην έκθεση και αυτό θα πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Πρόκειται για ελάχιστε προδιαγραφέ στι οποίε θα πρέπει να προσαρμοστούν τα κράτη-μέλη. Οι διάφορε πτυχέ είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσε. Εμεί οφείλουμε να καταφέρουμε να βρούμε τον τρόπο να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα, γιατί τα προβλήματα των στρεβλώσεων είναι γνωστά η δουλειά της ε, Task Force ε, θα πρέπει αυτά να τα λύσει και αυτή η οδηγία ε, τα επαναλαμβάνει όλα. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πόση δουλειά πρέπει να γίνει σε αυτή την Επιτροπή και εύχομαι μαζί με τη Μαριάν Μαγκίνες και τους συγκεκριώδες ηγητές να κάνουμε πραγματικά σημαντική δουλειά, να συμπληρώσουμε αυτή τη δεύτερη φάση μετά το Omnibus ώστε να καταστεί πιο διαφανής και ε, ισότιμη αυτές οι, οι δυνατότητες, αυτές οι πιθανότητες τρέβλωσης για όλους τους φορείς του τομέα. Και ελπίζω πως εδώ θα μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε και το θέμα της ε, στρέβλωσης για, τις, ε, για τα σήματα τα σήματα, τα εμπορικά, των μεγάλων ε, αλυσίδων που δημιουργεί πρόβλημα. Δημιουργεί πρόβλημα γιατί οι μεγάλες αλυσίδες ε, παράγουν τα δικά τους προϊόντα με το δικό τους σήμα ε, και έτσι στρεβλώνεται η κατάσταση και με τους παραγωγούς. Σας ευχαριστώ πολύ και ελπίζω να τα καταφέρουμε να προλάβουμε μέσα σε αυτή τη θητεία να ολοκληρώσουμε τη μελέτη αυτή της πρόταση. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Αρχίζουμε να πιστεύουμε τα θαύματα λέει ο, λέει ο Πρόεδρος, η κυρία Μαγκίνες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Φαντάζομαι πως η ατμόσφαιρα που επικρατεί εδώ αντικατοπλίζει το γεγονός ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι που βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο. Σας ευχαριστώ, με Επίτροπε, που τιμήσατε τη δέσμευσή σας στην ακρόασή σας ότι θα δουλεύατε και θα ε, κάνατε προτάσεις για αυτό το θέμα. Θέλω να αναφέρω τον συνάδελφο Νταντά, ε, που δεν μπορεί να είναι παρόν, αλλά θέλει και εκείνος να σας ευχαριστήσει και να σχολιάσει μαζί με μένα ότι φυσικά πρόκειται για ένα πρώτο βήμα και το Κοινοβούλιο Κοινοβούλιο θα δουλέψει σκληρά για να εξασφαλίσει πώς θα επιτύχουμε τους στόχους μας. Δεν είναι σήμερα η μέρα για τις λεπτομέρειες, γιατί είναι μέρα ορόσημο. Και πολλοί από εμά δεν συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικό είναι αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ καιρό πήρε να πείσουμε πολύ κόσμο ότι αυτό πρέπει να γίνει. Γιατί α το πούμε ξεκάθαρα, όταν πάει κανεί στο σούπερ μάρκετ φαίνονται όλα λαμπερά, καινούργια και τέλεια. Όλα είναι εκεί και μπορούμε να διαλέξουμε. Αυτό που κάνουμε σήμερα όμως είναι να ανοίξουμε το καπάκι στις ιστορίες που κρύβεται πίσω από την παροχή ολόκληρης αυτής της αλυσίδας. Οι δυσκολίες αυτών που δεν έχουν την εξουσία, δεν έχουν την επιλογή και δέχονται διαρκώς πίεση ως παραγωγή για να δώσουν αυτήν την λαμπρή ποιοτική τροφή στου Ευρωπαίου καταναλωτέ. Και πρέπει να ανοίξει το καπάκι αυτό αυτή τη ιστορία, γιατί δεν είναι πολύ ωραία αυτή η ιστορία. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη και να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής επίσης, τον Ζαν Κλοντ για τη δική του δέσμευση για λύσεις σε αυτό το θέμα. Θέλω επίση αν μου επιτρέπετε τρία δευτερόλεπτα, να μιλήσω για κάτι ευρύτερο. Είναι μια πρόταση που έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή. Έχουμε μια κοινή γεωργική πολιτική που θα μεταρρυθμιστεί και που υπόκειται σε δημοσιονομικέ πιέσει. Έχουμε γεωργού στη χώρα μου που αντιμετωπίζουν μια ακόμα κρίση λόγω άνευ προηγουμένου καιρικών συνθήκων που επικρατούν, σίγουρα έχουν επηρεαστεί από κλιματική αλλαγή. Έχουμε οικογένειε που αντιμετωπίζουν φοβερές πιέσεις αυτή τη στιγμή. Αν μπορείτε να το δείτε αυτό που σας δείχνω εδώ και σας το διαβάζω. Πρόκειται για μια ιστορία που δημοσιεύθηκε στον Ολλανδικό Τύπο αυτή την εβδομάδα. Η Ευρώπη θρέφεται από το αίμα 100 γεωργών κάθε χρόνο για, και θα σας το στείλω γιατί δεν έχουμε συλλογές, ε, συγγνώμη, στατιστικά στοιχεία για τους γεωργούς που πεθαίνουν, χάνουν τη ζωή τους στα αγροκτήματα. Ε, ένας, ε, γνωστό ειδικό ε, είπε στην, ε, στην Ιρλανδία πως αυτή είναι η ιστορία που κρύβεται πίσω από την αλληλετροφημική μας αλυσίδα. Ελπίζω πως ε, κάπως θα λογικευτούμε λοιπόν, θα σταματήσουμε αυτή την πίστευτη πίεση στους γεωργούς που αντιμετωπίζουν πιθανότητες ατυχήματος που χάνουν τη ζωή τους στη αγροκτήματά τους να έχουμε μια δίκαιη κατάσταση ειδικά για τους γεωργούς γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι δίκαιο το σύστημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κατάινεν. Η κυρία Κατάινεν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ Επιτρόπε και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα που κατέθεσε αυτή την πρόταση της πολύ σημαντικής αυτής οδηγίας, γιατί είναι το σωστό εργαλείο να αντιμετωπιστούν οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές στην ε, αλυσίδα των τροφίμων. Και το κοινοβούλιο μας και άλλα εθνικά κοινοβούλια Περίμεναν εδώ και καιρό. Και είναι σωστή η χρονική συγκυρία για να ενισχύσουμε την θέση των γεωργών. Τώρα θα πρέπει να γίνει αυτό. Τώρα που αναθεωρούμε και ανανεώνουμε και την ΚΑΠ. Είναι πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η πτύχη και θα επηρεάσει τον ε, προπολογισμό και θα επηρεάσει σημαντικά και τα, τον τρόπο ζωής ε, και λειτουργίας των αγροτών. Συμφωνώ σε ό,τι αφορά το θέμα της προστιθέμενης αξίας στην αγορά τροφίμων, στην αλυσίδα των τροφίμων. Το γεγονός ότι πολλά εθνικά κράτη-μέλη έχουν εθνική νομοθεσία για την ε, οδηγία πλαίσιο αυτή. Και θα ήθελα να τονίσω ότι στο σημείο αυτό η Ευρώπη και η νομοθεσία θα πρέπει να επιδείξουν επαρκή ευελιξία προκειμένου να εφαρμοστούν σε ε, εθνικό επίπεδο, γιατί δεν ε, χρειάζονται σε όλους τα ίδια μέτρα. Για παράδειγμα, στη Φιλανδία οι δύο πιο μεγάλοι χοντρικοί πολιτές έχουν 85% ε, του συνόλου της αγοράς. Τελευταίο στοιχείο που θα ήθελα να αναφέρω. Θα είναι σημαντικό να ενισχυθεί και η πτυχή της διαφάνειας σε ό,τι αφορά την διατροφική αλυσίδα και από πλευράς των καταναλωτών. Πιστεύω ότι ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πώς έχει κατανεμηθεί αυτή η προστιθέμενη αξία του τροφίμου που αγοράζει. Και να σας ρωτήσω, κύριε Επίτροπε, πώς θα βελτιωθεί αυτή η πτυχή της διαφάνειας στη διατροφική αλυσίδα στα πλαίσια της οδηγίας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ Θέλω καταρχάς να ε, Συγχαρώ και να ευχαριστήσω τον κύριο Πίτροπο Χόγκαν για αυτή την πρόταση που θέλει να ενισχύσει τη θέση των γεωργών στην ε, τροφιμική αλυσίδα και που ε, υποχρέωση πληρωμής εντός 30 ημερών των παραγωγών για συμφωνίες οι οποίες μονομερώς ε, αναστέλλονται. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ήδη να πω αυτός ο κανόνας και εύχομαι, ε, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ε, εξέταση αυτή τη πρόταση οδηγία να ολοκληρωθεί όσο γίνεται πιο σύντομα. Στην Ιταλία, για κάθε ευρώ που δαπανά ένα καταναλωτή, λιγότερο από τα 15 ε, λεπτά πάνε στον παραγωγό. Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούνται για την μεταποίηση και για την ε, διανομή. Με αυτή την πρόταση οδηγία αναγνωρίζεται επιτέλου ότι οι ανισορροπίε εισόδων τη τροφιμική αλυσίδα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με ε, κατεπηγόντω, ώστε να βελτιωθεί η διαπραγματευτική εμπορική ισχύ των γεωργών που είναι πραγματικά έρμε των εμπορικών πρακτικών και των μεγάλων εταιριών διανομής και των, μεγάλων σούπερ μάρκετ. Στην πρότασή μου του Union Act τον Ιούλιο του 2017 ήδη το ανέφερα. Πιστεύω πως είναι το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ανταγωνισμού θα πρέπει να συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο αποτελεσμα... μιας πιο αποτελεσματικής αγοράς αλλά για να το καταφέρει αυτό χρειάζεται περισσότερη διαφάνεια πάνω απ' όλα και καλύτερη ενημέρωση μέσα στο πλαίσιο της αλυσίδας προμηθειών καθώς και ενίσχυση των μέσων για την συλλογή πληροφοριών στην αγορά. Οι τιμές εντός της τροφιμικής αλυσίδας θα πρέπει να αντικατοπρίζουν καλύτερα την προστιθέμενη αξία των προτεραιών γενών παραγωγών. Ε, θα προσθέσω ότι κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο οι επαγγελματικέ οργανώσει ε, που θα πρέπει να φτιάξουν πλατφόρμες αλλά και να επιτραπεί έτσι στους γεωργούς να παρουσιάζουν και να υποβάλουν χωρίς φόβο καταγγελίες. Και άρα είναι Καλό νέο, καλό νέο είναι επίσης η συνεργασία που ζητά από το Κοινοβούλιο μας η Κομισιόν. Είναι αυτονόητη. Όλοι μαζί πρέπει να δουλέψουμε για να βελτιώσουμε τη θέση των Γεωργών. Ευχαριστώ. Η κυρία Αγγιλέρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι σημαντική μέρα σήμερα και θέλω να σας συγχαρώ, κύριε Επίτροπε, γιατί το έχουμε συζητήσει πολύ αυτό και έχουν περάσει επίτροποι και επίτροποι και κανένας δεν ε, μπόρεσε να μας υποβάλει μια οδηγία ή κάποια ρύθμιση για αυτή την υπόθεση. Πραγματικά και ειλικρινά, όπως και η κυρία Μαγκίνε, θεωρώ πως είναι ιστορική στιγμή, δεν είναι η στιγμή για τις λεπτομέρειες, αλλά είναι θεμελιώδη σημασία στο να μιλήσουμε για μια ε, οδηγία για τις αθέμετες πρακτικές. Δεν είναι εύκολο ε, και γι' αυτό θέλω πραγματικά ειλικρινά να σας ε, συγχαρώ. Δίνεται μια μεγάλη ελπίδα Καταρχάς, περισσότερα θα τα συζητήσουμε φυσικά δεν είναι όπω ένα κανονισμός, αλλά είναι μια καλή ε, πρόταση οδηγία για να προχωρήσουμε και είναι καλύτερο και από ό,τι ε, τι είχαμε μέχρι στιγμή. Θέλω να σας υποβάλω μια ερώτηση για την υπόθεση των ε, μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η πρότασή σας δεν μου φαίνεται κακή, αλλά θα ήθελα να καταλάβω ακριβώς γιατί ακριβώς εκεί τι αναφέρατε. Είναι καλή ιδέα και βέβαια θα πρέπει να συμπληρωθεί γιατί άλλο πρόβλημα είναι η πώληση με ζημία. Υπάρχει και ένα πρόβλημα και υπάρχει και απόφαση του δικαστηρίου για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και υπάρχει και ένα άλλο θέμα ότι δηλαδή τα μεγάλα σούπερ μάρκετ έχουν ένα τεράστιο βάρος ε, ε, και επιβάλλουν ε, τις προδιαγραφές. Όμως το ίδιο συμβαίνει και με τις μεγάλες βιομηχανίες. Και εσείς μιλήσατε για τη λακταλή, αναφερθήκατε στις λακταλίες ή άλλες μεγάλες εταιρείε που επίσης έχουν δυνατότητα επιβολής τιμών. Έχω επηρεάζουν τον καθορισμό των τιμών ε, που καταβάλλονται στους παραγωγούς. Ξεκινάμε λοιπόν με μια καλή αρχή για να λύσουμε το πραγματικό πρόβλημα των γεωργών. Το πραγματικό πρόβλημα των γεωργών είναι αυτό. Δεν μπορούμε να ξεχνάμε πως η μεγάλη βιομηχανία ασκεί τεράστια πίεση και ότι θα πρέπει και για αυτήν να συζητήσουμε στο μέλλον. Συγχαρητήρια και καλή επιτυχία στη συζήτηση. Η κυρία Χεράντζ Γκαρσία, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όπως ήδη είπε η κυρία Γιλέρ και η κυρία Μακίνες, θα πρέπει να σας συγχαρούμε. Πάνω από μια δεκαετία ζητάμε αυτή την πρόταση είναι μια μέρα γιορτή για μας ε, και σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ γιατί είναι πολύ θετικό βήμα. Είναι κάτι που ζητάνε οι γεωργοί, οι καταναλωτοί και εμείς εδώ και οι πολιτικοί αυτής εδώ της Επιτροπής. Πιστεύω, όπως το είπα και χτες, ότι υπάρχουν κάποια σημεία μετά από μια προσεκτική ανάγνωση ε, πρέπει να πούμε πως αυτό το έγγραφο που είναι καλό μπορεί να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο από εδώ, από τη δική μας Επιτροπή και εσείς ο ίδιος το αναγνωρίσατε. Ε, ένα από τα σημεία το τόνισε η κυρία Γκυλερά, που δεν χρειάζεται να το επαναλάβω, είναι το ρόλος των μεγάλων ε, επιχειρήσεων. Και αυτές ε, κάνουν αθέμητες πρακτικές, ακολουθούν μάλλον ε, αθέμητες πρακτικές. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε όλες ε, τις ε, πλευρές και όλους τους φορείς. Ξέρω πως είμαστε σε καλά χέρια με τον εισηγητή μας, ε, του έχω εμπιστοσύνη. Κάτι ακόμα που είναι πολύ ενδιαφέρον, στην Ισπανική νομοθεσία ας πούμε υπάρχει υποχρεωτική και ε, ε, υποχρεωτικά πρέπει οι συμβάσεις να γίνονται γραπτά και γι' αυτό μπορούμε κάπως να το βελτιώσουμε γιατί αυτό το γεγονό ότι είναι υποχρεωτικές οι γραπτές οι συμβάσεις αυτό έχει βελτιώσει πολύ την κατάσταση για τους παραγωγούς. Είναι ένας δρόμος αυτός που θα μπορούσαμε ίσως να ακολουθήσουμε. Είναι κρίμα που είναι οδηγία και όχι κανονισμός και αυτό πρέπει να το τονίσουμε γιατί έχουμε έτσι λιγότερη ισχύ και αν αφήσουμε τα κάτι μελη να ερμηνεύουν, αυτά οι δυνατότητε ερμηνείας αποδυναμώνουν το έγγραφο και την ε, διάταξη. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη του συνεταιρισμού. Είναι κάτι που θα είναι ενδιαφέρον να το έχουμε υπόψη, γιατί οι κανόνες, οι προδιαγραφές των ίδιων των συνεταιρισμών σε σχέση με του ίδιου του συνεταιριζόμενου, ε, ορίζονται μεταξύ του. Ε, ε, μέσα στο, σε κάθε συνεταιρισμό λοιπόν ε, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι ένα, μια πρόταση κλειδί στο εμπόριο, ε, στον αγροτροφημικό τομέα και θα προσπαθήσουμε και εμείς να δουλέψουμε να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο. Ο κύριος Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε εδώ και που μας ε, κάνατε αυτή την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Φυσικά, πολλοί συνάδελφοι και συμφωνώ μαζί τους καταγγέλνουν ότι το όλο θέμα του καρτέλ έχει αποτύχει, αλλά η ευρωπαϊκή ρύθμιση για τα καρτέλ είναι ουσιαστικά η εθνική ρύθμιση για τα καρτέλ σε ό,τι αφορά τα ολιγοπόλια, στις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ, τα οποία επιτράπηκαν. Άρα βλέπουμε πως αυτό καταπιέζει τις ε, υφιστάμενες αλυσίδες. Πιστεύω λοιπόν ότι η πρόταση είναι καλή και είμαι από ένα κράτος μέλος την Ιταλία όπου υπάρχουν ήδη τέτοιοι κανόνες ό,τι αφορά για παράδειγμα την προθεσμία 30 ημερών και το καθεξής και είχαν ε, πολλά θετικά πολλές θετικές επιδράσεις. Στην αρχή υπήρξε μεγάλη αντίδραση, αλλά στη συνέχεια είδαμε ότι λειτουργεί το σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν αυτό αποδεικνύει ότι κάποια μέτρα πρέπει να περνάνε. Και μάλιστα με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό που με ανησυχεί σε ό,τι αφορά τις αλυσίδες στο σούπερ μάρκετ είναι ότι όλο και πιο πολλοί αντικαθεστούν τον νομοθέτη και βγάζουν δικά τους ε, κανόνες σε ό,τι αφορά τους προμηθευτές για παράδειγμα και έτσι οι προμηθευτές βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να το σκεφτούμε αυτό. Επί της αρχής δεν είναι δυνατόν οι αλυσίδες μεγάλων σούπερ μάρκετ να παίζουν προς τα έξω τους καλούς και ευγενικού και να επιβάλλουν διάφορες υποτίθεται διατάξεις προστασίας και τελικά να δυσκολεύουν τη ζωή και να πατάνε τους ε, προμηθευτές. Αυτό λοιπόν είναι που θα πρέπει να κοιτάξουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι για την πρόταση. Η κυρία Πύρικα, σας ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω και τον Επίτροπο Όγκαν. Έχω μια συγκεκριμένη ερώτηση να κάνω. Εγώ προσωπικά θα προτιμούσα κανονισμό και όχι οδηγία. 20 χρόνια μας απασχολεί το θέμα αυτό. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Ο αγοραστής πληρώνει μέσα σε 30 ημέρες στην Ολλανδία και αυτό το έγραψε μια μεγάλη εφημερίδα ή τα σούπερ μάρκετ πληρώνουν μετά από 30, όχι 30 αλλά 60 ημερές οι τράπεζες, ελπίζω να με ακούτε επίτροπε τα φυλάν τα χρήματα αυτά και τα χρησιμοποιούν και στη συνέχεια ο υπουργό μας Μα δεν με ακούτε, επίτροπε, πολύ φοβάμαι. Την ακούσατε την ερώτησή μας. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Μία ερώτηση, η οποία τέθησε και στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο. Ρώτησε, λοιπόν, ζήτησε λοιπόν ε, ο συνάδελφός μου από τον Υπουργό να το επιλύσει το θέμα αυτό σε ό,τι αφορά τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα. Γιατί το θέμα αυτό μας απασχολεί εδώ και χρόνια και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους κάναμε το πρώτο βήμα. Αλλά είναι ένα πραγματικό βήμα το οποίο μπορούμε πραγματικά να υλοποιήσουμε. Πιστεύετε. Ευχαριστώ. mulțumesc foarte mult, Ευχαριστώ πάρα πολύ, ο κύριος Μπούτα. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Επίτροπο. Σας ευχαριστούμε για την πρόταση αυτή που μας υποβάλλατε. Όπως είπαν και οι συναδελφοί, είναι πολύ σημαντική χρονική συγκυρία για τους ε, αγρότες. Να πω το εξή με σαφήνεια, ότι οι αγρότες προφανώς πρέπει να βγάζουν ένα κέρδος. Αν δεν μπορούν να πολλούν τα προϊόντα τους με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάζουν ένα ελάχιστο κέρδος και να επιβιώσουν, εμάς θα εξαφανιστούν και τελικά θα έχουμε πιο ακριβά προϊόντα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σταθερότητα για τους αγρότες, να τους δώσουμε αυτή τη σταθερότητα σε ό,τι αφορά τώρα το εμπόριο σε όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γιατί στη Ρουμανία αντιμετωπίζουμε ένα σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη τιμή του γάλακτος, το γάλα, το καλοκαίρι, συγγνώμη. Πέφτουν οι τιμές σε σχέση με το χειμώνα. Και τελικά οι αγρότες να ξαναγκάζονται να πουλούν το γάλα τους για τιμή κάτω της ε, παραγωγή. Μα αυτό δεν θα του οδηγήσει να κλείσουν τελικά. Σε ό,τι αφορά την τιμή πώληση των προϊόντων, είναι τεράστιε οι διαφορές στις τιμές. από την ε, φάρμα μέχρι το ράφι του σούπερ μάρκετ. Και σε κάποιες περιπτώσεις ε, η τιμή του νερού είναι πιο υψηλή από την τιμή του γάλακτος. Μα αυτό θα πρέπει να το κοιτάξουν οι ενώσεις γεωργών. Είμαι από μια χώρα που αντιμετωπίζει έντονα τέτοια προβλήματα. Τέλος. Οι αγρότες και οι ενώσεις αυτές, οι συνεταιρισμοί θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να έχουν και δικά τους καταστήματα να πόλουν τα προϊόντα τους. Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί ένα καλό παράδειγμα για να μην εξαρτώνται τόσο πολύ οι συνεταιρισμοί και οι αγρότες από τα σούπερ μάρκετ. Um, Ευχαριστώ. Επιτέλους, μια καλή είδηση. Έχουμε μια νομοθετική πρόταση. Αλλά δεν είμαι πεπισμένος ότι κανένας μας ε, ότι εμείς θα μπορούσαμε τώρα δηλαδή να πούμε ειλικρινά στους ε, γεωργούς ότι τώρα επιτέλους θα πληρωθούν ε, τίμια για το προϊόν τους. Ε, χρειαζόμαστε ακόμη 2,5 χρόνια μέχρι να περάσει και να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία και θα έπρεπε να ενισχυθεί ούτως ή άλλως. Και γιατί να μην ξεκινήσουμε ανάποδα. Γιατί να μην προτείνουμε τις πιο ισχυρές προτάσεις και μετά οι συνομοθέτες αν θέλουν ενδεχομένω να αποδυναμώσουν κάπως το κείμενο. Γιατί, κοιτάξτε, οι πραγματικές αθέμητες εμπορικές πρακτικές που όλοι διαπιστώνουμε είναι ότι η γεωργία είναι επικεφαλής σχετικά μικρών επιχειρήσεων που πρέπει να αντιπαρατεθούν με μερικές από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου, είτε είναι μεταποιητές, είτε είναι εργοστάσια, είτε είναι αλυσίδες διανομής. Τι διαπραγματεύσει τώρα μπορεί να γίνει έτσι. Φυσικά ευνοούνται οι ισχυρότεροι. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε. Οι γεωργοί θα πρέπει τουλάχιστον να καλύπτουν το κόστος τους. Γιατί κανείς δεν μπορεί να υποχρεώσει τους αγοραστές όπως περιγράφονται εδώ να πληρώσουν μια σωστή τιμή που να ανταποκρίνεται στις, ε, στην κατάσταση της αγοράς, την οποία βέβαια μπορούν να ε, προσαρμόσουν εκείνο όπως θέλουν. Εδώ αναφέρονται οκτώ μέτρα που θα πρέπει να απαγορευτούν, αλλά τέσσερα από τα 8 επιτρέπονται αν αναφέρονται στο συμβόλαιο. Μα ακριβώ κατά τη διάρκεια διαπραγμάτευση για τη σύναψη συμβολέου ασκούν την ισχύ του και την υπεροχή του οι ισχυρότεροι. Άρα πρέπει να ενισχυθεί η πρόταση. Γιατί όπω σα είπα, οι γεωργοί σε μεγάλο βαθμό η επιβίωσή του εξαρτάται από αυτήν την πρόταση. Όσο ισχυρότεροι είναι, τόσο ισχυρότερη θα είναι και οι γεωργοί όταν πρέπει να διαπραγματευτούν με μερικέ από τι μεγαλύτερε εταιρείε στον κόσμο. Άρα αυτή τη στιγμή είναι άνισος ο ανταγωνισμός. Ο κύριος Γιάρ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ένας περίφημος φιλόσοφος. Είπε ότι οι φιλόσοφοι μέχρι τώρα ερμήνευαν τον κόσμο, αλλά το θέμα είναι να, τους αλλάξουμε, να τον αλλάξουμε. Τώρα λοιπόν κάνουμε μια προσπάθεια να αλλάξουμε κάτι έστω σε ένα βαθμό. Πού βλέπω τα προβλήματα. Πολλοί σας είναι χάρισαν. Εγώ πού βλέπω τα προβλήματα, πού πρέπει να προσέξουμε. Το σύστημα πρέπει να εφαρμοστεί αποτελεσματικά, όχι υπερβολικά γραφειοκρατικά. Κοιτάξτε, επί των εγγράφων όλα είναι άριστα. Αλλά να μην, σκεφτάμε, να μην ξεχνάμε ότι στη μέση όλων αυτών είναι το εισόδημα του γεωργού, η εκμετάλλευση. Πρέπει να βρούμε ένα σύστημα που να είναι αποτελεσματικό, όχι απλώς ε, στο τέλος απλώς τα σούπερ μάρκετ να συμπληρώνουν άλλα τρία έντυπα και να λένε ότι όλα είναι άψογα. Πρέπει λοιπόν να μην υπάρξει υπερβολική γραφειοκρατία, να είμαστε αποτελεσματικοί δεν θέλουμε, αυτό το λέω συχνά, να βελτιώσουμε τις στατιστικές αλλά την πραγματικότητα. Λοιπόν, είχατε το θάρρος όμως να υποβάλλετε αυτή την πρόταση, επιβάλλατε στην Κομισιόν να περάσει και θα έχετε και την πλήρη στήριξή μας για την εφαρμογή της. Κοχάου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλημέρα. Επίτροπε, εγώ συμμερίζομαι κάποιες από τις προτάσεις ε, που, κάναν, ε, που κάνατε κύριε Επίτροπε και οι συνάδελφοι για τη χρήση όμως της οδηγίας και, του, και όχι κανονισμού είναι μακρύς χρόνοι αλλά δεν μπορούν να δώσουν απαιτήσεις ε, στις τρέχουσες κρίσεις όπως αυτή στην περιφέρειά μου της Σικελίας στην περιφέρειά μου της Σικελίας όπου γνωρίζετε ότι η κατάσταση των Γεωργών είναι δραματική. Οι συγκελοί Γεωργοί ε, δεν ε, μπορούν να σταθούν στην, στην ανταγωνισμό, υπάρχουν αθέμετες εμπορικές ε, πρακτικές, οι μεγάλοι εταιρείε διανομής τους έχουν πιέσει. Σε τρία χρόνια δεν θα προλάβουμε να τους βοηθήσουμε αν καθυστερήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι νωρίτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Ριμπέρο. Ευχαριστώ. Πρόκειται για μέτρα πολύ εκτεμένα και πολύ αναμενόμενα για τους γεωργούς. Εμείς εργαζόμαστε για να προστατεύσουμε τους γεωργούς που είναι το πιο αδύναμο σχολικό σε αυτή την αλυσίδα ε, την τροφιμική. Θέλουμε να κάνουμε κάποια βήματα για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους μικρούς κυρίως γεωργούς που είναι πολύ σημαντικό για ε, πολλές περιφέρειες ε, ε, που υστερούν. Θα πρέπει να δούμε όμως και τις λεπτομέρειες. Μας υποβάλλατε μια οδηγία ε, με συγκεκριμένους προσανατολισμούς και συγκεκριμένες ρυθμίσεις από την πλευρά την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ο ορισμός των εμπορικών πρακτικών είναι σημαντικός και είναι σημαντικό επίσης να έχουμε και την ανωνυμία στις καταγγελίες. Αυτό είναι οι σημαντικές προτάσεις. Θα πρέπει επίσης να μπορούμε να συνάπτουμε συμβάσεις που θα επιτρέπουν τη σταθερότητα για τους γεωργούς και, και η αρχή που θα επιβάλλει τις κυρώσεις, ποια θα είναι, πώς θα εφαρμόζονται και πώς αυτές οι αρχές ε, θα συνεργάζονται με τις δικαστικές αρχές κάθε κράτος μέλος. Ε, τέλος, να πω και εγώ ότι πρόκειται για ιστορική μέρα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σίγουρα θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να έχουμε μια αποτελεσματική οδηγία και οι γεωργοί μας να είναι ικανοποιημένοι για να επιτύχουμε έναν από τους στόχους που ξεκινήσαμε στη, αυτή τη θητεία. Κύριος Σταραμπέλα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, όντως η πρόταση οδηγίες είναι πολύ καλή. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, οι γεωργοί είναι οι μόνοι ανεξάρτητοι επαγγελματίε που μπορούν να πουλούν με ζημία. Γενικά απαγορεύεται. Αλλά οι γεωργοί όχι μόνο δεν μπορούν να καθορίσουν την τιμή στην οποία θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, αλλά σήμερα πολλοί πουλούν με ζημιά. Δουλεύουν με ζημία. Θα πρέπει λοιπόν η ουσία του νομοθετήματος αυτού θα πρέπει, θα πρέπει να είναι λοιπόν ότι θα πρέπει να απαγορεύεται να πουλάνε κάτω του κόστου στο μέλλον. Και δεύτερον, Παράλληλα, μέσω άλλων μέτρων και στην μελλοντική κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να επανέλθουμε σε μηχανισμούς ρύθμισης των αγορών, ούτως ώστε οι τιμές να είναι πιο αξιοπρεπείς, τουλάχιστον να φέρουν κάποιο κέρδος. Να αποφύγουμε, να αποφύγουμε αυτές τις απαράδεκτες, ιδιαίτερα για τους νέους γεωργούς διακυμάνσεις που διστάζουν να επενδύσουν στην γεωργία γιατί δεν βλέπω προπτικές, ενώ οι κίνδυνοι είναι πανταχού παρόντες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το κατάλογο των ομιλητών. Δεν βλέπω κανέναν άλλο συνάδελφο. Α, η κυρία Πετήρ. Κυρία Πετήρ. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Ευχαριστώ για την πρότασή σας. Και ευχαριστώ και την κυρία Μαγκίνες πρώτα απ' όλα, η οποία ασχολήθηκε με το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι σκόπιμη αυτή η πρόταση. και να σταματήσουν αυτές οι αθέμητες πρακτικές. Γιατί η γεωργοί υφίσταται τις συνέπειες. Όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, νομίζω ότι υπάρχει συστηματική παραβίαση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πληρωμές. Το διαπίστωσα στην ε, Κροατία. Δεν γίνεται σεβαστή η προθεσμία των 30 ημερών Πολλές φορές ε, πληρώνονται οι γεωργοί έξι μήνες μετά. Και γίνονται και άλλου τύπου παραβιάσεις. Τελευταία στιγμή, για παράδειγμα, τα προϊόντα τους τους επιστρέφονται. Και δεν ναι, ξέρουν ούτε καν πού να τα βάλουν. Δεν έχουν χώρους αποθήκευσης. Είναι λοιπόν ε, ιδιαίτερα θετική αυτή η πρόταση. Ναι, μεν είναι οδηγία. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα καλό παράδειγμα για να δείξουμε ότι σε ενωσιακό επίπεδο ε, κάνουμε κάτι για να καταπολεμηθούν οι μαύρες ή γκρίζες πρακτικές. Να δείξουμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους γεωργούς, τα προϊόντα τους, το μέλλον τους. Ο κύριος Φαντεκάνδελαρα, ευχαριστώ πάρα πολύ πρόεδρε και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος ότι, γιατί υπάρχει μια συμφωνία για την βασική αντιμετώπιση της πρότασης του Επιτρόπου. Η επιθυμία να στρεχθούν οι αγρότες και να καθοριστούν σωστές πρακτικές. Θα πρέπει, θα ήθελα και εγώ να έχουν περιληφθεί και άλλα στοιχεία, αλλά εν πάση περιπτώσει αποτελεί μια βάση κίνησης. Θα ήθελα να μας εκτιμήσετε τον αντίκτυπο της πρότασής για τους παράγοντες που είναι πριν από τον αγρότη, τραπέζες, ε, παραγωγούς ε, ζωοτροφών κτλ. Πώς θα επηρεάσει λοιπόν αυτή η πρόταση αυτούς που βρίσκονται πριν από τον Γεωργό στην αλυσίδα παραγωγής. Okay, Ωραία. Λοιπόν, τώρα πραγματικά μίλησαν όλοι όσοι ήθελαν να μιλήσουν. Λοιπόν, είχα και μία μυστική ερώτηση. Πόσοι πρόλαβαν να διαβάσουν το κείμενο της οδηγίας. Αλλά ο Επίτροπος ε, βλέπει ότι έχει διάφορες σελίδες με σημειώσεις, οπότε να του δώσω το λόγο. Να ξαναπώ ότι φυσικά δεν είναι πανάκια αυτή η πρόταση. Δεν θα βελτιωθεί εντυπωσιακά και αμέσως η κατάσταση των Γεωργών. Δεν γίνεται αυτό με ένα μέτρο για τις αγορές των προϊόντων, αλλά είναι ένα τμήμα της ε, στρατηγικής τριών ε, μέτρων που θέλουμε να υιοθετήσουμε. Το πρώτο ήταν ε, με τη βοήθεια του κυρίου Ντεκάστρο και του κυρίου Αντέ και των άλλων σκιωδών και όλων των συναδέλφων τη Επιτροπή εδώ και την ισχυρή σα στήριξη. Κάναμε λοιπόν αυτό το πρώτο βήμα για τι οργανώσει των παραγωγών. Και πάντα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα μέσω τη μεταρρύθμιση τη ΚΑΠΑΓΑΜΑΠΗ. Δεύτερον, έχουμε λοιπόν αυτό το νομοθέτημα για τις αθέμητε πρακτικέ που το προσπαθούμε να το προωθήσουμε 19 χρόνια. Και φυσικά μπορούμε να βελτιώσουμε και το πεδίο εφαρμογή. Αυτό είναι θέμα των συνομοθετών. Και συμφωνώ απόλυτα ότι υπάρχουν κάποια θέματα. Τα αναφέρατε. Δεν καλύπτονται όλα. Ιδιαίτερα ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Βαν Κίντελαρ. Για παράδειγμα, αυτή η... δεν καλύπτονται τα θέματα των ε, προμηθευτών ε, λεπασμάτων και άλλων εισρώων, αλλά ε, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Είναι λοιπόν μια προσέγγιση ελαχίστων προδιαγραφών. Και γιατί προτείνουμε οδηγία. Θέλουμε να βελτιώσουμε αυτά που ήδη υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Να βελτιώσουμε την πρωτοβουλία για την αλυσίδα προμηθειών. Γιατί αν δεν ήταν πρόβλημα δεν θα χρειαζόταν να λάβουν μέτρα 20 κράτη-μέλη. Δεν θα έχει υπάρξει αυτή η πρωτοβουλία που είναι βεβαίω εθελούσια. Και υπάρχει εδώ και 7 χρόνια. δεν υπήρχε πρόβλημα δεν θα υπήρχαν όλα αυτά. Και όλοι Εκτό από του γεωργού βέβαια, συμμετέχουν σε αυτή την πρωτοβουλία για την αλυσίδα προμηθειών. Ελπίζω η σημερινή μα αναγγελία να επιτρέψει και στου παραγωγού παραγωγούς βεβαίως να συμμετάσχουν, να πάψουν αναποκλεισμένοι σε αυτή την πρωτοβουλία. Και πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι στην αλυσίδα για να βρούμε λύσει. Θα υπάρξει νομοθεσία, αλλά θα υπάρχουν και οι δυνατότητες τα κρατημέλη να κάνουν περισσότερα, αν θέλουν να σχεδιάσουν σωστά το σύστημα εφαρμογής νομοθεσίας, να καθορίσουν την εποπτική αρχή και αυτές οι εποπτικές αρχές με την πρωτοβουλία μας θα συντονίζονται. Ευχαριστώ όλους ε, τους συναδέλφους για τη γενική προσέγγιση με την οποία συμφωνούν, αλλά φυσικά και πάλι τονίζω, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν σημεία όπου θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε την πρόταση. Και γι' αυτό πιστεύω ότι θα συνεργαστούν ε, στενά οι τρει θεσμοί. Βεβαίω η κυρία Μαγκίνε έχει δίκιο. Πολλέ πιέσει υφίστανται οι Γεωργοί. Πρέπει να δουλεύουν ανεξάρτητα από τον καιρό. Πρέπει να θρέψουν τις οικογένειές τους, πρέπει να πληρώσουν τα δάνειά τους. Και φυσικά αισθάνονται μεγάλη πίεση. Έχουν θέματα ασφάλειας, έχουν θέματα ψυχικής υγείας. Αλλά Ελπίζω. Βεβαίω η πρότασή μα ε, έχει περιορισμένο πεδίο εφαρμογή, αλλά ελπίζω να επιτρέψει ιδιαίτερα στου μικρότερου παραγωγού να αποκτήσουν λίγο περισσότερη εμπιστοσύνη στη δουλειά του. Για τη Φιλανδία. Γνωρίζω τα προβλήματα, ότι υπάρχει πολύ υψηλή συγκέντρωση στην αγορά. Αλλά αυτό είναι θέμα που πρέπει να επιλύσουν τα κράτη-μέλη. 85% είναι βέβαια πολύ ψηλό ποσοστό συγκέντρωση. Αυτό δεν είναι καλό για τον καταναλωτή. Γενικότερα για τη λειτουργία της αγοράς. Το είπε και η κυρία Κατάινεν. Η κυρία Αγγιλέρα και η κυρία Εράνθ αναφέρθηκαν στους μικρούς γεωργούς. Βεβαίω εστιάζουμε σε αυτούς. Γιατί πολλές φορές είναι αδύναμη θέση του. Οι μικρομεσαίες Ακόμη και εάν ε, ε, ε, είναι ιδιοκτησία γεωργών, μπορούν παρόλα αυτά να είναι η μάντα μετάδοση των αθεμήτων πρακτικών μέχρι τον πιο αδύνατο κρίκο που είναι ο Γεωργό όπω ξέρουμε. Αυτό προσπαθούμε να αποφύγουμε. Αυτή είναι η λογική τη πρότασή μα. Για τα γραπτά συμβόλαια. Έχουμε τέσσερι τέτοιε πρακτικέ που τι έχουμε εντοπίσει. Είπαμε ότι υπάρχουν άλλε τέσσερι που μπορεί να ε, αξιοποιηθούν ως αθέμητες πρακτικές αν δεν υπάρχει συμφωνία. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία για αυτές τις τέσσερις για να μπορέσουν να ισχύσουν. Για την εμπορία και την διαφήμιση δηλαδή, τα παρόμοια θέματα. Ο κύριος Καπούτο, όπως και πολλοί άλλοι, αναφέρθηκε στο πώς θα εφαρμοστεί η οδηγία και ο κύριος Γιάρ. Ε, άμα αυτό είναι ζωτική σημασία, η εφαρμογή και ο έλεγχος εφαρμογής. Βεβαίως θα συνεργαστούμε για να το καταλάβουν τα κρατη θα, παρακολουθήσουμε πολύ στενά ποιες είναι αυτές οι εποπτικές αρχές και πώς θα λειτουργήσουν. Γιατί βεβαίως ε, απομακρυνόμεθα από τη φιλοσοφία ότι ε, ένα ταυτόσιμο μέτρο ισχύει παντού και μπορεί να λύσει ε, όλα τα προβλήματα. Όχι, βασιζόμαστε πολύ περισσότερο στην επικουρικότητα. Θέλουμε να υπάρχουν και αναλογικές κυρώσεις εάν υπάρξουν προβλήματα, εάν ε, εξακολουθούν να υφίστανται αυτές οι πρακτικές. Αλλά το βασικό είναι να ενισχυθεί η διαπραγματευτική θέση των γεωργών και να εντοπίζονται πολύ σύντομα οι καταγγελίες, ιδιαίτερα οι ανώνυμες. Αυτό είναι σημαντικό και για τις δύο πλευρές. Αν κάποιος κάνει ένα ισχυρισμό, και δεν αντιμετωπιστεί σύντομα, τότε μπορεί η φήμη, ε, για παράδειγμα, ε, του αγοραστή να φύγει. Θέλουμε να βασιστούμε σε αυτά που γίνονται στην Ισπανία και στον Ηνωμένο Βασίλειο για να προχωρήσουμε. Και συμπεριλαμβάνονται και τα υποχρεωτικά συμβόλαια, βεβαίω. Βεβαίω, συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογή. Και οι, συνεργατικέ ενώσει, οι συνεταιρισμοί συμπεριλαμβάνονται. Γιατί ξέρουμε πολύ συχνά ότι οι συνεταιρισμοί εισάγουν τους δικούς τους εσωτερικούς κανόνες. Θα τους λάβουμε υπόψη. Εάν μέσω αυτών των εσωτερικών κανόνων των συνεταιρισμών μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα του γεωργούς, βεβαίως. Βεβαίως. Γιατί όχι, να υπάρξει οδηγία στον τομέα αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Ο κύριος Ντόρφμαν αναφέρθηκε στους κανόνες που πρέπει να ισχύουν για τις αλυσίδες διανομής. Ναι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην ε, σπατάλη τροφίμων. Θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Η κυρία Πύρικα αναφέρθηκε σε ένα θέμα στην Ολλανδία. Να ασχοληθούμε καλύτερα με το θέμα αυτό μέσω του συστήματος για τις ε, καθυστερημένες πληρωμές. Γιατί υπάρχει στην πρότασή μας η απαγόρευση των καθυστερημένων πληρωμών. Υπάρχει ένα θέμα βέβαια, ξέρω, στο Ολλανδικό Κοινοβούλιο και ίσως θα μπορούσατε να μας δώσετε στοιχεία. Ο κύριος ε, Μπούντα αναφέρθηκε σε αυτά που είπε ο πρόεδρος Γιούνκερ. Ήταν μια ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον Πρόεδρο που εξασφάλισε το θέμα αυτό να είναι υψηλή προτεραιότητας. Γιατί όταν ένα θέμα είναι προτεραιότητας φυσικά ε, πρέπει να ε, αναλυφθεί δράση γι' αυτό. Και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γιατί το, το, το συμπεριέλαβε στο πρόγραμμά του 2017 μας επέτρεψε να υποβάλουμε αυτέ τι προτάσεις. Κύριε Κάθη, Δεν κατάλαβα τι εννοείται. Δηλαδή θα διατυπώσουμε αρχικά μια ε, πολύ στεναρή πρόταση η οποία κατόπιν θα αποδυναμωθεί. Είπατε ξεκινήστε με την ε, πιο ισχυρή πρόταση ώστε κατόπιν να την αποδυναμώσουμε. Αυτό δεν είπατε. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων. Νομίζω ότι το να ξεκινάει κανείς με πολύ ισχυρή θέση και τελικά να την αποδυναμώνει, ξέρετε ότι όπως και στη συμφωνία της ε, Μεγάλης Παρασκευής ε, αντίστροφη είναι η διαδικασία. Ξεκινά από μια πιο ε, μετριοπαθή πρόταση και μετά προσπαθεί να την ενισχύσει. Αλλά, αλλά σε έξι μήνε καταφέραμε κάτι να κάνουμε γι' αυτό. Αντιστρέψαμε την κατάσταση. Ελπίζω κάτι να κάνετε, γιατί νομίζω ότι και το Κοινοβούλιο συμμετείχε στην ε, Διοργανική Συμφωνία για τι ε, καλύτερε ρυθμίσει. Ίσως καμιά φορά δεν καταλαβαίνετε τι στηρίζετε. Ανέφερα τον κύριο Γιάρ. Ναι, Θέλουμε να υπάρχουν ε, οι αναγκαίες εκθέσεις. Διαχείριση των κινδύνων και δίκτυα ασφαλείας. Βεβαίως, το αντιμετωπίζουμε και θα υπάρξουν περαιτέρω προτάσεις. Και οι νέοι γεωργοί βεβαίως πρέπει να ενισχυθούν ιδιαίτερα. Ελπίζουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα για να βοηθήσουμε τους νέους να παραμείνουν στη γεωργία ή να ξεκινήσουν στα διαδρομή στη γεωργία. Ελπίζω να μην ξέχασα κανένα. Δεν έχω καμία πρόθεση. Η κυρία Πετήρ Αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα εφαρμογή στα κράτη-μέλη. Συμφωνώ απόλυτα. απόλυτα. Ο κύριος Κοράου ανάφερε διάφορα σημαντικά θέματα. Ο κύριος Μακάρθη. Α, σας, ε, εκνεύρισα. Δεν ξέρω τώρα εάν η ε, στρεβλώνεται αυτό που είπα ή δεν καταλάβατε. Είπα, γιατί να μην ξεκινήσετε με τις πιο ισχυρές διατάξεις για να, για να προστατεύσετε τους γεωργού από αυτέ τι αθέμητε, να αγωνιστείτε για να ε, ισχύσει αυτό, ενώ εσείς ξεκινάτε από μια πιο αδύναμη ε, διατύπωση και ζητάτε οι συνομοθέτε να την ενισχύσουν. Μα το κάνω για να σας δώσω και κάτι να κάνετε κι εσείς, λέει ο κ. Χόγκαν. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορώ να έχω όλε τι απαντήσει ευθύ εξ αρχής. Πρέπει να περάσω και από την Επιτροπή αυτέ τι πρότασει. Εσεί πρέπει να περάσετε τι ιδέες σα από το Κοινοβούλιο. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ο καθένα ε, αγωνίζεται για αυτό που πιστεύει και προσπαθεί να επιτύχει ό,τι μπορεί. Εγώ υπέβαλα μια πρόταση την πρώτη οποτεδήποτε. Ευχαριστώ λοιπόν για τη στήριξή σας και θα δούμε και τις ε, τροπολογίες σας. Ο κύριος Κοράου αναφέρθηκε σε διάφορα θέματα ανταγωνισμού, θέματα στη Σικελία, Ξέρω ότι τώρα στην Ιταλία είναι πολύ ιδιαίτερη η πολιτική κατάσταση. Μπορείτε να υποβάλλετε διάφορες προτάσεις. Και ίσω αν έχετε σημαντικά αξιώματα στο μέλλον να μπορέσετε να εφαρμόσετε πολλέ από αυτέ τι ιδέε. Αλλά θα πρέπει βεβαίω τότε να υπάρξει στήριξη, να κερδίσετε την υποστήριξη και από άλλε πολιτικέ ομάδε και τάσει, όπω και εγώ στην Επιτροπή, αλλά εντοπίσατε μια σειρά από σημαντικά θέματα που θα μπορούσαμε να εντάξουμε στο πεδίο εφαρμογή αυτή της πρότασης. Οπότε, και τέλο, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ του ε, συνεργάτε μου από την DG Agri που είναι παρόντες. Έκαναν τεράστια δουλειά, άκουσαν τι απόψει, σα, ε, διατύπωσαν προτάσει, συνεργάστηκαν με άλλε γενικέ διευθύνσει και δεν ήταν εύκολο. Και όπω θα διαπιστώσει και ο κύριο Κάρθη στο μέλλον, όταν θα εξετάσουμε αυτή την πρόταση, το βασικό είναι να πείσετε, να, να ε, παρουσιάσετε τα επιχειρήματά σας και να πείσετε. Αλλά σε κάθε φάση εμείς ε, προτείνουμε ό,τι ισχυρότερο μπορούμε. Και εγώ και οι συνεργάτες μου, οι υπάλληλοι μου. Κοιτάξτε, κανείς δεν πρέπει να φοβηθεί την εφαρμογή αυτής της πρότασης εάν δεν κάνει κάτι αθέμητο. Προσπαθούμε να καταργήσουμε τις αθέμητες πρακτικές και θέλουμε ισότιμες συνθήκες συνεργασίας μεταξύ όλων όσων συμμετέχουν στην ε, αλυσίδα παραγωγής και εμπορίας τροφίμων. Άρα, εάν είστε σωστός, δεν πρέπει να φοβηθείτε τίποτα από τις προτάσεις μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Επίτροπε. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι. Και να έχετε υπόψη σας παρακαλώ ότι ο Επίτροπος ε, θα πρέπει να... Μάλλον, ε, η πρόταση του Επιτρόπου για την οδηγία έπρεπε να περάσει και από τους άλλους Επιτρόπους. Και οι γενικοί διευθυντές έπρεπε να συνομιλήσουν και να συμφωνήσουν. Και κατά δεύτερον, Χρειαζόμαστε και πραγματικό διάλογο στην ε, αλυσίδα παραγωγής και προμήθειας, γιατί έχω την εντύπωση ότι όλοι μιλούν στα πλαίσια των πολιτικών τους ομάδων και θα θυμάστε ότι είχε γίνει και ένα κίνημα κατά της πρόσκλησης ε, παραγόντων από την αλυσίδα παραγωγή. Χωρί ουσιαστικό διάλογο όμω δεν πρόκειται να υπάρξει αποτέλεσμα. Γι' αυτό λοιπόν απευθύνω έκκληση για την εξαγωγή τέτοιου διαλόγου στην αλυσίδα παραγωγή. Με τον τρόπο αυτό θα καταστεί δυνατόν να σημειωθεί πραγματική πρόοδο. Δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει απαραίτητα συμφωνία. Αλλά πάντα χρειάζεται να γίνεται διάλογος. σίγουρα θα παρουσιαστούν και σημεία διαφωνίας, αλλά θα βρούμε σίγουρα και τρόπους να μην τηρήσουν τη διαταξή της οδηγίας σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τα συμβόλαια, τις συμβάσεις και το τι επιτρέπεται από αυτές. να ευχηθούμε στην εισηγήτρια και στους κοιόδης ε, κάθε επιτυχία στις εργασίες τους. Να πάνε καλά και ομαλά οι εργασίες αυτές. Η ομάδα μας θα είναι ιδιαίτερως ισχυρή. Και μπορούμε να υπολογίζουμε στην καλή θέληση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου και σε ό,τι αφορά την Omnibus. Ελπίζουμε λοιπόν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον Επίτροπο και όλους τους συναδέλφους. Την άλλη εβδομάδα έχουμε συνάντηση στο Στρασβούργο χωρίς την Επιτροπή. Και σας ευχαριστώ και πέρα στις